Good morning. Uh, we'll start the meeting now. Uh, Καλημέρα σας. Να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Έχουμε στη διάθεσή μας όλες τις γλώσσες σήμερα, εκτός από τα κροατικά. Η Άγνες, με. Ακούστε με, είναι σήμερα τα γενέθλιά της, της Άγνες, αν τη δείτε αργότερα. Ίσως να μην είναι τώρα εδώ γιατί είναι γιορτάζει. Να σας πω ότι σύμφωνα με τον κανονισμό η μετάφραση των τροπολογιών στην Επιτροπή δεν θα γίνεται στα, προς τα κροατικά, αυτό προς γνώση σας μόνο και έπειτα επίσης προς ενημέρωσή σας ε, να σας πω ότι έχουμε μια ομάδα επισκεπτών. Το Ευρωκοινοβούλιο και το γραφείο ενημέρωση του Κοινοβουλίου στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει καλέσει 40 φοιτητέ ε, δημοσιογραφίες από το Πανεπιστήμιο του Λίτζ για να παρακολουθήσουν αυτή τη συνεδρίαση της Επιτροπής Απασχόλησης στη διάρκεια των ψηφοφοριών. Και η κυρία Κούνεβα έχει καλέσει μια ομάδα επισκεπτών 21 ατόμων που θα είναι εδώ ανάμεσα στις 11 και στις 12.30 σήμερα. Οπότε έχουμε κόσμο που θα μας ακούει όχι μόνο μπροστά στις τηλεοπτικές οθόνες, αλλά και μέσα στην ίδια την αίθουσα της συνεδρίασης. Σημείο 3 της ημερήσιας έταξης που αφορά τα πρακτικά μπορούν να εγκριθούν χωρίς αλλαγές. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Ευχαριστώ. Τέταρτο σημείο ετήσια έκθεση για το 2013 για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και θα δώσω το λόγο αμέσως στον εισηγητή Τάβιτ Κάσα από το ΕΛΚ. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης Κάποιοι από τους πιο σημαντικούς ε, παράγοντες ήταν ε, ότι πρόκειται για το πρώτο ε, σχέδιο. Όπως γνωρίζετε, στο πρώτο σχέδιο περιοριζόμαστε σε συγκεκριμένο αριθμό λέξεων, αλλά ελπίζω πως πολλά θα προσθεθούν μέχρι ότου να συζητήσουμε το τελικό σχέδιο. Ιδιαίτερα όσον αφορά την μείωση ε, της ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, αυτό είναι πολύ ευπρόσδεκτο και είναι πολύ ευπρόσδεκτο ότι υπάρχει αύξηση των θέσεων απασχόλησης. Τα στοιχεία δεν είναι απαραίτητα θετικά για όλα τα κρατημέλη, αλλά υπάρχει μια θετική Ανοδική τάση και αυτό είναι καλό νέο. Συμφωνώ με τη σύσταση της ΕΚΤ ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην εφαρμογή των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίασης που είναι φιλικά προς την ανάπτυξη. Ε, όσον αφορά τώρα τον κανονισμό περί θεσμικού πλαισίου για την Οικονομική Νομισματική Ένωση, καλωσορίζω την έκκληση της ΕΚΤ να βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί αυτός. Όμως ο συντονισμός μέτρων και οικονομικών μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να προχωρήσουν από κοινού ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτή είναι μια πολύ σύντομη έκθεση που έχω και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Προσβλέπω στις ε, τροπολογίες και στις συμβολές σας που θα γίνουν από εδώ και μπρος. Ευχαριστώ κύριε Κάζα και δίνω το λόγο στην, στον... στο Χάβι Λόπες. Uh, ε, Mr. Lopez is not here. Είναι εδώ ο κύριος Λόπες. Then I'll give the floor to uh, uh, Ulrike Trebesius from the ECO. Ulrike Trebesius από τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Ούτε αυτή είναι εδώ. Περιμένουμε κανέναν. Η φιλελεύθερη τότε, η κυρία Χάρκιν. Εσείς εδώ είστε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και να ευχαριστήσω και τον ε, συντάκτη της γνωμοδότησης. Δυστυχώς ε, όταν ε, μιλούσε, μιλούσα με κάποιον άλλον, αλλά την έχω διαβάσει και συνεργάστηκα και με τον κύριο Γκάς επί του θέματος. Ένα-δύο σχόλια ε, από την έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την οποία πρέπει να ομολογήσω ότι μια ματιά της έριξα μόνο, δεν τη διάβασα αναλυτικά, Ε, θεωρώ ότι η γνωμοδότηση του κυρίου Κάσα είναι μάλλον ε, υπερβολικά θετική. Ναι, μεν ε, πρέπει να είμαστε θετικοί, αλλά κάπου αναφέρεται στη μείωση του ποσοστού ανεργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2010 μέχρι το 2013 και ναι, μεν είναι σωστό αυτό, αλλά αν δείτε τα στοιχεία του 2012 θα διαπιστώσετε ότι δυστυχώς υπάρχει αύξηση στην ανεργία για το τελευταίο έτος. Επομένως, ίσως θα έπρεπε λίγο να ισορροπήσουμε τα πράγματα στη γνωμοδότηση από αυτού. Επίσης, ε, να σχολιάσω και την παράγραφο 5, στην οποία ε, καλωσορίζει την έκκληση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προς τα κράτη-μέλη για να ε, εφαρμόσουν συγκεκριμένα μέτρα, κυρίως για τη βελτίωση της ευελιξίας. Δεν υπάρχει τίποτα κακό με την ευελιξία, αλλά αν μόνο αυτό έχει το σχόλιο εδώ για τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, ναι μεν, αλλά μπορούμε να εξετάσουμε και άλλα θέματα για τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας. Επίσης θα πρέπει να πούμε και κάτι για την ε, ανεργία των νέων σίγουρα. Αυτά. Έχω και ένα-δυο άλλα πράγματα. Αλλά σε γενικέ γραμμέ θεωρώ πολύ καλή τη γνωμοδότηση και θα υποβάλω κάποιε τροπολογίε και είμαι βέβαιη ότι θα συνεργαστούμε πολύ καλά επί του ζητήματο. Thank you. Uh, I'll now try with the uh, madam. Ευχαριστώ. Να προσπαθήσουμε. Να προσπαθήσουμε τώρα με Δεν ξέρω αν θέλετε, έχετε το λόγο. Ε, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ε, εξέτασα το σχέδιο αυτό και υπάρχουν κάποια ερωτήματα τα οποία προκύπτουν. Καταρχάς, θα ήθελα να ξέρω Από πού βγήκε αυτό το 20,8%. Γιατί μιλάμε για μια μεγάλη μείωση των ανέργων. Δεν το βλέπω αυτό πώς προκύπτει βάσει των στοιχείων της Eurostat. Ύστερα θα ήθελα να ξέρω τι εννοούμε με έναν προϋπολογισμό ε, φιλικό προς τον προϋπολογισμό. Δεν έχουμε ούτε καλό προϋπολογισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε την ανάπτυξη που θέλουμε. Και υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία θεωρώ ότι δεν είναι καθόλου προβληματικά, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να πω ότι επιφυλάσσουμε γιατί θα καταθέσουμε κάποιες τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. I'll give the floor to... Ευχαριστώ και θα δώσω το λόγο στον κύριο Ιαρίκ από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους, ε, το συνάδελφο για τη γνωμοδότησή του, αλλά όπως και ο προκάτοχός μου, μάλλον η προλαλήσασα, να σας πω ότι μου δημιουργεί αρκετά προβλήματα. Καταρχάς, κανείς δεν διαπιστώνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μείωση της ανεργίας και μάλιστα τόσο μεγάλη. Νομίζω ότι είναι το αντίθετο από αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Επίσης, το σημείο 3 όταν συζητούμε τις ε, ε, προκλήσεις ε, της δημοσιονομικής εξυγίανσης με στόχο την ανάπτυξη, όλοι γνωρίζουν αυτή τη στιγμή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζει να βιώνει μία έναν αποπληθωρισμό με όλες τις συνέπειες που μπορεί να υπάρχουν και για τους πολίτες. Και στο σημείο και 4 και 5, όπου για άλλη μια φορά μας ε, ενημερώνεται ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να υποστηρίξει τις μεγάλες πολιτικές μεταρρυθμίσεις όπως έχουν αποφασιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μας λέτε ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις αφορούν την αγορά εργασίας, την αύξηση της ευελιξίας, ε, τη βελτιστοποίηση των συνθήκων που θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν απασχόληση, όλος ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι όλοι αυτοί οι όροι που χρησιμοποιούνται είναι οι όροι της αποτυχίας του σήμερα. Και επομένω, εγώ δεν θεωρώ ότι μπορούμε να εγκρίνουμε ένα τέτοιο προσανατολισμό και μάλιστα ως μονόδρομο χωρίς να υπάρχει και καμία ε, ένσταση. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε. Παραδείγματο χάρη γιατί δεν τίθεται το ερώτημα ε, του πώς ε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική ε, ε, Τράπεζα παίζει συνεχώς ένα παιχνίδι με την Ομισματική Ένωση για τις τράπεζες χωρίς αυτό να βοηθά σε οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, κατά την άποψή μου, προβλήματα τα οποία τίθενται από τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση και προτείνω να επαληθεύσουμε καταρχάς τα στοιχεία. Και όσον αφορά τις συστάσεις, τις οποίες υποτίθεται ότι θα πρέπει να προσυπογράψουμε κι εμείς, ε, εγώ δεν μπορώ να τις ε, προσυπογράψω και γι' αυτό ακριβώς και θα καταθέσουμε και σχετικές τροπολογίες. Ε, νομίζω ότι δύσκολα όμως θα συμφωνήσουμε. Καρή Μαντελή από τους Πρασίνους. Oh, πριν δώσω το λόγο στου υπολείπου, να δώσω και το λόγο στην κυρία Λάουρα Άτζια. Καλημέρα, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχουμε κάποιες παρατηρήσεις για το σχέδιο γνωμοδότησης του συναδέλφου Κάζα. Για το σημείο 1, έστω ότι σε μία μακροοικονομική κατάσταση στην οποία γίνεται ένας γενικότερος υπολογισμός του πώς θα μπορούσε να είχε προχωρήσει ε, η ανεργία τα τελευταία τρία χρόνια ε, Παρ' όλα αυτά πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένε ιδιαίτερε περιπτώσει, παραδείγματο χάρη ε, η περίπτωση τη χώρα μου, τη Ιταλία, που ε, είναι εντελώ αντίθετη προ τι προβλέψει αυτέ. Θεωρούμε λοιπόν ότι δεν είναι δυνατόν να θεωρήσουμε ότι έχουμε μείωση του ποσοστού τη ανεργία. Θα πρέπει σίγουρα να αναφερθούμε και στην κατάσταση που αντιμετωπίζει το κάθε κράτο μέλο και σε καμία περίπτωση η κατάσταση αυτή δεν αντανακλά ε, μείωση. Όσον αφορά το δεύτερο σημείο, μια ερώτηση. Γιατί αναφερόμαστε σε αύξηση της μισθολογικής δαπάνης ε, όταν δεν αναφερόμαστε σε όλα τα κράτη-μέλη και ε, αναφερόμαστε μόνο σε αυτά που είναι εκτός της Ευρωζώνης. Μήπως θα έπρεπε να έχουμε και τα στοιχεία για τα ε, κράτη-μέλη εντός της Ευρωζώνης. Επίσης, πώς μπορούμε να έχουμε και πάλι ανάπτυξη και να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας σεβόμενοι τους όρους του ε, προϋπολογισμού που είναι πραγματικά μέγενοι για τους μικρούς επιχειρηματίες και την πραγματική οικονομία. Κατά την άποψή μας είναι αδύνατο να θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνονται σεβαστές κάποιες δεσμεύσεις ε, που ε, είναι ουσιαστικά τιμωρία γιατί δεν επιτρέπουν σε καμία περίπτωση να έχουμε ανάπτυξη. Πώς μπορούμε αυτά λοιπόν να τα συμφιλιώσουμε με τη διάθεση της ανάκαμψης. Για το σημείο 5 η σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη μεταρρύθμιση στην αγορά εργασίας και τη μεγαλύτερη ευελιξία. Ε, εδώ να σας πω ότι ο μόνος τρόπος να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας και να δώσουμε ανάκαμψη στην οικονομία είναι μια δραστική μείωση στην ομογενοποίηση των φορολογικών πολιτικών, ε, να υπάρχουν μεγάλες εισρωές χρημάτων ε, στις τράπεζες, γιατί αν τα τράπε... οι τράπεζες κατά κάποιο τρόπο μπορούσαν να δώσουν και δάνεια στους μικρούς επιχειρηματίες, θα μπορούσαμε να το αντιληφθούμε. Αλλά επειδή τα χρήματα τα οποία δίνονται στις τράπεζες ε, δίνονται αποκλειστικά και μόνο για κερδοσκοπία, ε, θεωρούμε ότι είναι περιττό να τους δίνουμε και άλλα χρήματα. Και επίσης να σας πω Eh, Κάτι για το σημείο αυτό. Η έρευνα του ευρωσυστήματος σχετικά με την περιουσία και την κατανάλωση των οικοκυριών, ναι, είναι σημαντική, διότι είναι σημαντικό να διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει πλέον περιουσία για κατανάλωση στα νοικοκυριά, κυρίως στη χώρα μου, στην οποία πραγματικά ε, έχουμε πλήρη αποπληθωρισμό και ε, οι περιουσίες έχουν ε, μειωθεί δραστικά και δυστυχώς είναι τα πρώτα πράγματα που οι άνθρωποι αναγκάζονται να ξεπουλήσουν για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Ευχαριστώ. Thank you. Ε, then I'll Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στον Σον Σαν. Ευχαριστώ. Για την παράγραφο στο σημείο 5 να πω ότι δεν χρειαζόμαστε περισσότερη ευελιξία. Δεν υπάρχει πρόβλημα με την ευελιξία στην αγορά εργασία. Το κομμάτι τη αγορά εργασία όπου υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία ακριβώ είναι εκείνο το κομμάτι τη αγορά εργασία όπου έχει και τη λιγότερη δουλειά. Όλη η ευελιξία επικεντρώνεται ανάμεσα στους νεότερους, ε, τους ανθρώπους που έχουν τις λιγότερες δεξιότητες, τις γυναίκες, ε, τους ε, μερικώς απασχολούμενους, τους απασχολούμενους από γραφεία interim. Εκεί που υπάρχει λοιπόν η περισσότερη ευελίξια υπάρχει και η περισσότερη χρόνια μαζική ανεργία. Και το δίδαγμα που πρέπει να αποκομίσουμε είναι ότι δεν, όχι ότι χρειαζόμαστε περισσότερη ευελιξία, αλλά ότι Ευελιξία σημαίνει εκμετάλλευση στην ουσία. Δεν είναι αυτή η απάντηση για την απασχόληση στο χαμηλότερο, ε, στο χαμηλότερο κομμάτι της αγοράς εργασίας. Αυτό που θέλουμε είναι δουλειά, ε, δουλειές, ε, δεξιότητες και βασικά τα προβλήματα αγοράς είναι προβλήματα ζήτησης από την οικονομία που προκαλούνται από τις πολιτικές λιτότητας που ασκούνται τα τελευταία χρόνια. Οπότε παρακαλώ όλοι όσοι ενδιαφερόμαστε για αυτά τα θέματα να μην ε, γοητευτούμε από την τσίχλα αυτή της ευελιξίας ε, χωρίς να σκεφτούμε τι σημαίνει πραγματικά και αν κάποτε θα προσέξουμε το γεγονός ότι δεν, δεν λειτουργεί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στον κύριο Ντομινίκ Μαρτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ να ευχαριστήσω καταρχήν τον εισηγητή που έκανε αυτές τις προτάσεις και να μιλήσω αμέσως μετά από αυτό που είπε ο τελευταίος ομιλητής πάνω στο σημείο 5 λέγοντας ότι η ευελιξία δεν δημιουργεί την απασχόληση αλλά την ανεργία. Δεν ξέρω για ποια χώρα μιλά αλλά στη Γαλλία πολύ, πολύ δεσμευτική νόμη, ο κώδικας ο εργασίας ε, ε, υποχρεώνει τις επιχειρήσεις στο κατόφ, σε κατόφλια δηλαδή πάνω από 10 ή πάνω από 50 εργαζόμενους ε, διστάζουν να προσλάβουν με συμβόλαια συμβάσεις αορίστου χρόνου αλλά ε, προσλαμβάνουν κόσμο με ε, συμβάσεις σε προσωρινού χρόνου. Στη Γαλλία μεγαλύτερη ευελιξία θα ήταν απαραίτητη. Τώρα η μείωση λέει της ανεργίας εδώ σε τέτοιο τεράστιο ποσοστό είναι απίστευτη. Ε, σίγουρα δεν συμβαίνει στη Γαλλία. Αλλά ίσως αυτή η ένδειξη να οφείλεται στην αύξηση της μερικής επισφαλούς εργασίας. Για το σημείο 2 βλέπουμε ότι η... Ε, ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να γνωρίζουμε περισσότερο τι συμβαίνει στην Ευρωζώνη. Αλλά σίγουρα είναι μια μεγαλειώδη ομολογία που λέει ότι όσο λιγότερο εργαζόμαστε με το ευρώ, τόσο περισσότερο ευημερούμε. Ε, δηλαδή, Αντίθετα, ο, αντίστροφα, όσο περισσότερο επιβάλλεται το ευρώ, τόσο περισσότερο αυξάνεται η δυστυχία και η επισφάλεια. Διαπιστώνουμε επίσης ότι ο στόχος 2020 με την λιτότητα και την δημοσιονομική εξυγένση έχει δημιουργηθεί προκληθή ανεργία. Τώρα, λέει ο Επίτροπος ότι με αυτό το πακέτο, το δημοσιονομικό, την λιτότητα ακόμα, θα δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης. Δυστυχώς όμως εδώ και 10 χρόνια βλέπουμε ότι ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Σημείο 4 λέει διαπιστώνει ο, τις προσπάθειες της ΕΚΤ για την βελτίωση του θεσμικού πλαισίου κτλ. και σημειώνει μια απώλεια επικυριαρχίας για τα κράτη-μέλη. Ε, εμείς φυσικά δεν είμαστε υπέρα αυτής της συστηματικής μεταφοράς ε, κυριαρχίας προς τις Βρυξέλλες. Το 5 ήδη το συζήτησα, το 6 ε, ανησυχούμε και για το 7 συνεχίζουμε να διερωτώμεθα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φουντούλης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, όσον αφορά την παράγραφο 1 για τη μείωση του ποσοστού ανεργίας δεν νομίζω ότι αντικατοπρίζει την πραγματικότητα. Τα πραγματικά στοιχεία δείχνουν ότι τα ποσοστά ανεργίας αυξάνονται δραματικά. Ειδικά μετά την καταιγίδα των φορολογικών βαρών που επιβάλλουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε ορισμένες χώρες όπως η Ελλάδα, τις οδηγούν σε κλείσιμο με αποτέλεσμα να χάνονται οι ήδη υπάρχουσες θέσεις εργασίας θα έπρεπε να γίνει προσπάθεια για τη διάσωση των ήδη υπαρχουσών θέσεων και εν συνεχεία να συμβάλλουμε ώστε να δημιουργηθούν και νέε θέσει. Στην παράγραφο 5, όταν λέμε ευελιξία, θα πρέπει να προσέξουμε ούτω ώστε να μην παρεξηγηθεί η έννοια με την έννοια τη εκμετάλλευση, μειώσει μισθών με λίγε ώρε απασχόληση εκ μέρου των εργοδοτών που απασχολούν του εργαζομένου κατά το δοκούν σημαίνει εκμετάλλευση. Στην παράγραφο 2, γιατί περιορίζουμε την αύξηση της μισθολογικής δαπάνης εκτός ζώνης του ευρώ. Γιατί στην πραγματικότητα στα κράτη-μέλη εντός της ζώνης υφιστάμεθα μείωση της δαπάνης, το οποίο στην πραγματικότητα σημαίνει μείωση μισθών, μείωση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων. Σας ευχαριστώ. Euh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν για τα γαλλικά, το γαλλικό ζήτημα γιατί ανεφέρθη. Μπορεί όμως να γίνει μια τελείως διαφορετική ανάλυση. Είμαστε μόνη χώρα που έχουμε 150.000 ανθρώπους επιπλέον που μπαίνουν στην αγορά ε, κάθε χρόνο χάρη σε μια δυναμική δημογραφία. Ε, εμείς χρειάζεται να δημιουργήσουμε λοιπόν ε, θέσεις απασχόλησης και βλέπουμε ότι η ανεργία αυξήθηκε τη στιγμή που έπαψε η ανάπτυξη και η ασφάλεια υπάρξει, υπάρχει μαζικά γιατί οι περισσότερες θέσει που δημιουργούνται είναι επισφαλού χαρακτήρα. Δεν μπορούμε να πούμε λοιπόν σήμερα ότι ε, τα, οι συμβάσει είναι ευνοικέ και ευνοούν την, ε, δηλαδή την, ε, αυτές ευνοούν την ανεργία. Τώρα, σε υπάρχει ακόμα ένα πολύ σημαντικό θέμα όσον αφορά το ανεργία. Προσοχή στις ε, στατιστικές δυσκολίες και στις στατιστικές ε, μεταμφιέσεις, γιατί η μείωση της ανεργίας ε, υπολογίζεται με βάση τις θέσεις απασχόλησης που είναι επισφαλής μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου, που στην ουσία μιλάμε για φτωχούς εργαζόμενους που δεν είναι πια άνεργοι, ναι, έχουν πλήρη απασχόληση και τότε μπορούμε όντω να πούμε ότι είναι μείωση της ανεργίας, αλλά στην ουσία πρόκειται για μια επέκταση της απασχόλησης κακής ποιότητας ε, αύξηση μάλλον της απασχόλησης κακής ποιότητας. Και κάτι ακόμα, η ΕΚΤ αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα. Χρειάζεται να χρησιμοποιήσει μια γλώσσα που λέει ότι ναι, χρειάζονται ε, φιλελεύθερες και διαστατικές αλλαγές. Αυτό δημιουργεί θέσεις απασχόλησης και ανάπτυξη. Είναι σχεδόν υποχρεωμένη να χρησιμοποιεί αυτή τη γλώσσα, αλλά και η ίδια δεν τα πιστεύει και πολύ πια αυτά που λέει. Και όταν ακούμε ο κύριο Ντράγκη που λέει ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι δηλαδή αν δεν υπάρχει δραστήρια δημοσιονομική πολιτική, κυρίω από την πλευρά των χωρών που το μπορούν αυτό, η, η, η, η ρευστότητα που εγώ η ΕΚΤ βάζω στην αγορά, δηλαδή το χρήμα που τυπώνω, δεν βρίσκει ε, ε, παραλήπτη γιατί δεν υπάρχουν επενδυτέ. Αυτό δεν χρησιμεύει σε τίποτα. Χρειάζεται διδαστήρια δημοσιονομική πολιτική και αυτό μας παραπέμπει στο μακροοικονομικό ζήτημα του σχεδίου των 300 δι κτλ. κτλ αλλά και εθνική δραστήρια δημοσιονομική πολιτική που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν βρίσκω λοιπόν την, ε, αυτά όλα στην έκθεση που μας ε, έχει δοθεί και επίσης θα πρέπει να μιλήσουμε για τη σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στην πολιτική διαχείριση και την ΕΚΤ. Ξέρω πως αυτή τη στιγμή αυτό δεν γίνεται, αλλά ίσως πρέπει να διαρωτηθούμε μήπως πρέπει να αλλάξουμε τις συνθήκες για αυτό το θέμα. Thank you, Madame Ribeiro. Σας ευχαριστώ κυρία Ριμπέιρο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ έχω κάποιες σημειώσεις που θα ήθελα να σας κοινοποιήσω σε σχέση με αυτή την έκθεση. Καταρχήν, αυτή η ανάλυση μου φαίνεται πως είναι εξαιρετικά ρόδινη και δεν ε, είναι προσαρμοσμένη και δεν αντικατοπτρίζει μάλλον τη γενική αίσθηση των Ευρωπαίων πολιτών. Ιδιαίτερα στην Πορτογαλία εμείς είχαμε πολύ αρνητική κατάσταση σε σχέση με το είδος της απασχόλησης που υπάρχει και που προσφέρεται και γι' αυτό θα θέλαμε να παρουσιάσουμε, να, μάλλον να επιστήσουμε την προσοχή για αυτή την έκθεση. Εν γέννη, Μιλάμε για πολύ επισφαλείς θέσεις επασχόλησης, μικρής ε, διάρκειας, πρόκειται για, στά, για είδη στάζ. Και εδώ ε, ε, μπορεί να υπάρξει μια εξέλιξη σε σχέση με την απασχόληση, αλλά πρέπει να δημιουργηθούν οι απαραίτητε προποθέσει για να έχουμε ποιοτική απασχόληση. Και παρά αυτού του δείκτε που εν γέννη ε, είναι πραγματικά θετικοί, θα πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή ότι σε ορισμένα κράτη-μέλη, ε, συμπεριλαμβανομένου του δικού μου, υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία όσον αφορά την απασχόληση, γιατί είναι τελείω επισφαλή η κατάσταση. Αυτό πρέπει λοιπόν να αναφερθεί γιατί σε κάποιες ε, χώρες πρέπει να γίνουν θετικές προσπάθειες ώστε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ποιοτικέ θέσεις απασχόλησης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θέλει κανείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει λόγο, να κάνει σχόλια. Αν όχι... Ο κύριος Κάζα θέλει να πάρει το λόγο. Καταρχάς, να πούμε ότι πρόκειται για μια έκθεση όπου μπορούμε να κάνουμε μια περιορισμένη γνωμοδότηση. Δεν μπορούμε να βάλουμε όλα όσα θέλουμε να πούμε. Προφανώς παρόλα αυτά. Πρέπει να παρουσιάσουμε μία έκθεση όσο το δυνατόν πιο ισορροπημένη. Συμφωνώ με την πλειοψηφία των συναδέλφων. Που μιλούν για θέματα δημιουργία τη συνεργασίε και το πόσο προσεκτικοί θα πρέπει να είμαστε όταν κάνουμε τέτοιε δηλώσει. Όταν αναφέρουμε δηλαδή θέσει ε, επισφαλή, θα πρέπει να δείχνουμε ιδιαίτερη προσοχή γιατί η έκθεση της ΕΚΤ δεν αναφέρεται σε τέτοιου είδους απασχόληση και σε θέσεις μερικής απασχόλησης. Θα συνεργαστώ στενά με τους συναδέλφους από τις διάφορες πολιτικές ομάδες και θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μια ισορροπή έκθεση προκειμένου να αποτυπώνονται οι σε όλου του κόσμου. Ευχαριστώ, λέει η, Πρόεδρο, η Πρόεδρος. 6 ε, Νοεμβρίου η προθεσμία για τις τροπολογίες στην Επιτροπή Επασχόλησης. Θα ψηφίσουμε 1η 2η Δεκεμβρίου στην Ίκον στις 8 Δεκεμβρίου και μετά θα περάσει στην Ολομέλεια του Φεβρουαρίου το θέμα αυτό του χρόνου. Σας ευχαριστώ. Και πάμε τώρα στο επόμενο, στην επόμενη γνωμοδότηση, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ετήσια έκθεση 2013. Και τώρα θα δώσω το λόγο για δεύτερη φορά στον κύριο Ντέιβιτ Κάζα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και πάλι, όπως για την γνωμοδότηση για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έχουμε τον ίδιο περιορισμό σε ό,τι αφορά την έκθεση της γνωματότησης. Προσπάθησα λοιπόν να περιοριστώ προκειμένου να υπάρξει και μια ισόρροπη αποτύπωση των απόψεων. Προωθεί λοιπόν τις ικανότητες και τα προσόντα των νέων η έκθεση. Αυτό είναι καλό. Λοιπόν. Όλοι ξέρουμε ότι χρειάζονται τέτοιες, ε, τέτοια προσόντα στην αγορά των εργασίας. Η επένδυση λοιπόν στους ε, νέους είναι ένας πολύ καλός τρόπος να προλάβουμε τις προκλήσεις ε, για το μέλλον. Ένα δισεκατομμύριο, για παράδειγμα, έχει δαπανίσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στον κλάδο αυτό. Για να είμαστε ανταγωνιστικοί, πρέπει να κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε και να υποστηρίξουμε την καινοτομία. Η καινοτομία, ωστόσο, μπορεί να είναι επικίνδυνη για τους επιχειρηματίες που εμπλέκονται στην διαδικασία αυτή και θα πρέπει να υποστηριχθούν. Και εδώ πιστεύω ότι θα πρέπει να προβλέπονται χρηματοδοτικές δυνατότητες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με υψηλό προφίλ κινδύνου. Επίσης, να υποστηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με επιπλέον χρηματοδότηση. Είναι θετικό ότι η Τράπεζα Επενδύσεων έχει αυξήσει κατά 50% σε σχέση με το 2012 την χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων γιατί δημιουργούν θέσεις εργασίας. Θα πρέπει να συνεχίσει η τάση αυτή. Σε ό,τι αφορά τώρα την ε, αξιολόγηση τριών πυλώνων, καλό την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να δώσει σημασία στους εξής ε, κριτήρια. Ποιότητα της ε, απασχόλησης και να δώσει σημασία στην απασχόληση ως την πύλη για μια βιώσιμη Ευρώπη. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να τονίζουμε το θέμα της ε, απασχόλησης των νέων και λοιπόν υποστηρίζω την απόφαση της Τράπεζας Επενδύσεων να υποστηρίξει την πρωτοβουλία για την νεολαία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και προσβλέπω στα σχόλιά σας και στις τροπολογίες σας. Ευχαριστώ. Thank you. Uh, σας ευχαριστώ. Ο κύριος Λόπες είναι εδώ από την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Όχι. Ο Ρίκε Τρεμπέσιος από την ε, ομάδα του ECR. μάλιστα, παίρνετε το λόγο για το ECR. Μάλιστα, πολύ ωραία. Ε, ε, ε, Σα ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να τα αξιολογήσω όλα αυτά με ένα θετικό τρόπο και θα ήθελα λοιπόν να πω ότι συμμερίζομαι την θετική εντύπωση του εισηγητή σε ό,τι αφορά τη χρηματοδομική δέσμευση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα προγράμματα υποστήριξης της νεολαίας. Εξίσου θετικά ξεολόγω, όπως και ο εισηγητής άλλωστε, τα θέματα των μέσων μικροχρηματοδότησης για την καταπολέμηση της, ε, του κοινωνικού αποκλεισμού. Και Ιδιαίτερο θα ήθελα να υπογραμμίσω δε το εξή στοιχείο. Η τράπεζα από το 2013, τουλάχιστον αυτό προκύπτει από την έκθεση, εξετάζει και προσεγγίζει εξατομικευμένα πλέον τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε κράτος μέλος, κατά ανάγκη δηλαδή, κατά περίπτωση. Για παράδειγμα, το μέσο της εγγύησης πιστώσεων για την Ελλάδα και την Κύπρο, Κύπρο, τέτοια, τέτοιες πιστώσεις για μικρές επιχειρήσεις όλα, αυτά, επιχειρήσεις, όλα αυτά είναι θετικές στάσεις που μπορούν να βοηθήσουν για την βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και της οικονομικής συγκυρίας στις χώρες αυτές, με τα διαφορετικά αυτά λοιπόν χρηματοοικονομικά μέσα. Στην έκθεση λοιπόν αναφέρεται και η επένδυση για τους νέους, για τα προσόντα των νέων, η προώθηση της κινητικότητας. Όλα αυτά είναι θετικά στοιχεία, θεωρώ. Με κάποια επιφύλαξη, την οποία άλλωστε πολλές φορές έχει παρουσιάσει το Κοινοβούλιο και σε ό,τι αφορά την ακρόαση για την ενεργεία των νέων, σημειώνουμε ότι η κινητικότητα σήμερα είναι κάτι το οποίο γίνεται αντιληπτό ως κάτι αρνητικό. Εφημισμός για, την, ε, για τον διωγμό των νέων από τη χώρα τους, από την πατρίδα τους, λόγω της οικονομικής κρίσης. Μία άλλη παρατηρήση τώρα. Σε ό,τι αφορά τα θέματα συγχρηματοδότησης που αναφέρονται για θέματα έργων για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Αυτό που θα ήταν σημαντικό είναι σε τέτοια έργα να λαμβάνονται υπόψη ε, και οι παραδοσιακές πηγές παραγωγής ενέργειας της κάθε χώρας και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας της ενέργειας. Κατά τα άλλα, θα καταθέσουμε σχετικέ τροπολογίε για να κάνουμε και περαιτέρω παρατηρήσει. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Στάινρουκ από το, την ομάδα των Σοσιαλιστών και των Δημοκρατών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχά, η έκθεση αυτή δεν είναι απόλυτα ταυτισμένη με την προηγούμενη έκθεση. Θεωρούμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τονίζονται καλά, αλλά θεωρούμε ότι θα πρέπει να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογή, να μην περιοριζόμαστε μόνο σε μικρομεσαίε επιχειρήσει όπω ορίζονται. Σημαντικό είναι επίση η προώθηση των προσόντων και των ικανοτήτων των ε, νέων. Πολύ σημαντικά προγράμματα αυτά, όπως και τα προγράμματα κατά του κοινωνικού αποκλεισμού είναι πάρα πολύ σημαντικά. Χρειαζόμαστε επίσης επενδύσεις στην εκπαίδευση, κατάρτιση, καινοτομία και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και θα καταθέσουμε λοιπόν σχετικές τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. I'll give the floor to Madam Harkin. Ευχαριστώ κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Για τη γνωμοδότηση αυτή νομίζω ότι μπορώ να συμφωνήσω με τον κύριο Κάσα που έχει πάλι και πιο θετικό ε, τόνο, συμφωνώ πλήρω μάλιστα, νομίζω ότι έχουμε μια καλή γνωμοδότηση εδώ και ένα-δυο παρατηρήσεις τι οποίε θα ήθελα να τονίσω εν συντομία. Ε, νομίζω ότι εκεί που αναφέρεται στη δέσμευση του Αντιπρόεδρου Κατάινεν ε, για να κάνει έκκληση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να γίνουν περισσότερες επενδύσεις ε, στην παιδεία, αυτό θα ήταν σημαντικό και στους νέους. Επίσης, ε, για τη δυνατότητα των μικροπιστώσεων, αυτή η δυνατότητα είναι κατά του κοινωνικού αποκλεισμού των ευάλωτων ομάδων και ε, το 2013 είχαμε 26 τέτοιες ε, συναλλαγές. Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία διότι ε, για όσους ήταν εδώ και την προηγούμενη φοιτεία θα γνωρίζετε ότι δώσαμε μάχη προκειμένου να υπάρξει αυτή η δυνατότητα. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προσπαθούν να έχουν μια προσέγγιση η οποία θα εξετάζει τις ανάγκες της κάθε κράτους μέλους. Και το γεγονός ότι επικεντρώνονται λίγο περισσότερο ε, στα λεγόμενα μεσαία ανώτατα όρια, ναι, ε, μιλάμε συνεχώς για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, αλλά έχουμε και ε, τις επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους που έχουν μεταξύ 250 και 500 υπαλλήλων και καλό είναι που η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επικεντρώνεται και σε αυτές τις επιχειρήσεις. Θα υπάρξουν κάποιες τροπολογίες από πλευρά μας, αλλά σε γενικές γραμμές ε, είναι θετική η στάση μας και μπορούμε να υποστηρίξουμε τα περισσότερα όπως αναφέρονται. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος από την Ενωτική Ιεροστερά που θα ήθελε να λάβει το λόγο. Όχι από ό,τι βλέπω. Η Καρή Μαντελή μέρος των Πρασίνων και πάλι δεν είναι εδώ. Η κυρία Άντζεα Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Παρά το γεγονός ότι είναι το ότι μπορεί να συνεισφέρει στην οικονομία η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα θέλαμε να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις. Αυτή τη στιγμή τα αποτελέσματα μέχρι τώρα μας φαίνονται ότι δεν είναι ιδιαίτερα καλά, διότι ο μηχανισμός αυτός ενεργοποιήθηκε σε μια στιγμή στην οποία η κρίση είχε ήδη φτάσει σε πολύ προχωρημένο επίπεδο και επομένως ε, πλέον ήταν προφανείς οι ζημίες. Το να δημιουργήσουμε συστήματα ε, βελτίωσης και ε, να βάλουμε ένα φρένο ήταν τελικά πάρα πολύ δύσκολο. Ακόμα και αν θεωρείται λοιπόν αποτελεσματικό μέσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι πρόκειται για ένα μέσο το οποίο ενεργοποιήθηκε μάλλον κατόπιν εορτής. και παρά το γεγονός ότι έχουμε πέντε χρόνια που εφαρμόζεται το μέτρο, δεν φαίνονται ακόμα προφανώς αποτελέσματα. Κάτι ακόμα το οποίο θα θέλαμε να σχολιάσουμε είναι όντω ότι είναι σημαντικό να γίνουν επενδύσεις στους νέους, αλλά η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα πρέπει να επενδύσει ε, μόνο όταν δεν δίνει τόσο μεγάλη ε, έμφαση στην ε, διατήρηση ε, της ε, βαθμολογίας στα 3α, αλλά τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει στους νέους. Αυτό δηλαδή που θέλουμε να επισημάνουμε είναι ότι ορισμένες φορές δεν είναι τόσο σημαντικό να έχουμε πρότυπα και απόδοσης πάρα πολύ καλά, αλλά το να παρέχουμε τα κατάλληλα μέσα ώστε να έχουμε αύξηση στην απασχόληση, κυρίως για τους νέους, και να επενδύσουμε στους ίδιους τους νέους. Και τέλος θα ήθελα να τονίσω κάτι το οποίο είναι κατά βάση αφορά Ιταλικό, αφορά την Ιταλία. Στην Ιταλία αυτοί οι οποίοι υποφελήθηκαν από αυτές τις επενδύσεις ήταν οι μεγάλες πολυεθνικές ε, στον ενεργειακό τομέα και στον τομέα των ε, υποδομών, ένα 35% ε, έλαβαν επενδύσεις από εκεί και είχαμε 10% για τη βιομηχανία, την ανάπτυξη και την έρευνα. Αν κάνουμε λοιπόν υπολογισμούς, ε, βλέπουμε ότι οι μικροί ε, και μεσαίοι επιχειρηματίες, που είναι αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε να υποφοληθούν περισσότερο από αυτές τις επενδύσεις, διότι αυτό αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Ιταλικής οικονομίας, ελάχιστα υποφελήθηκαν από αυτό το μέσο, γι' αυτό ακριβώς θα θέλαμε να καταθήσουμε και σχετικές τροπολογίες. Ευχαριστώ. Thank you. I'll give the floor to Mr. Ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στον κύριο Μαν. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξ ονόματος των σοσιαλιστών η κυρία Στάινμπρουκ είπε ότι οι μικρομεσές δεν αρκούν. Εγώ δεν συμφωνώ. Εγώ είμαι ευχαριστημένος που μπορέσαμε να σταματήσουμε ε, μάλλον να λάβουμε μέτρα ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων γιατί αυτές ε, είναι αυτές που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης. Γι' αυτό και είμαι ευτυχής που έχει φτιαχτεί ένα σύστημα διαβούλευσης μπορέσαμε να κλιμακώσουμε την παρέμβασή μας σε σχέση με τις ανάγκες του κάθε κράτους μέλους. Κάποιες μικρές επιχειρήσεις στη χώρα μου μπορεί να είναι μεγάλες σε κάποια άλλη χώρα. Πρέπει λοιπόν να μπορούμε να προσαρμοστούμε στις καταστάσεις και να εκτιμήσουμε κάθε φορά τις ευαισθησίες και τις επιχειρηματικές δομές. Πιστεύω πως αυτή, αυτή η η διαδικασία είναι σωστή και είμαι ευτυχή που η ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει λειτουργήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Η έκθεση αυτή αφορά, ο απολογισμό αφορά το 2013, ε, ο απολογισμό είναι εξαιρετικός, αυξήθηκε δε και ο εισηγητή το υπογράμμισε. Ε, τώρα, κινητικότητα μπορεί να είναι δίκοπο μαχαίρι πολλές φορές σημαίνει η ε, επένδυση χρημάτων για να μπορέσει ο κόσμος να μετακινηθεί. Αλλά η μετακίνηση μπορεί να είναι και μια ευκαιρία γιατί επιτρέπει να εργαστεί κανείς αλλού, σε άλλον τομέα ε, και μπορεί αυτό να μην μπορεί να το καταφέρει χωρίς ένα μικρό σπρόξιμο. Δεν είναι αρνητικό αυτό το σύστημα. Δεν θέλουμε να εισάγουμε συστηματικό την ομαδική ζωή, απλώς θέλουμε να μπορεί ο κόσμος να μετακινείται πιο εύκολα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτως ή άλλως πολλοί νέοι ήδη σκέφτονται πιο πέρα από τα εθνικά τους σύνορα. Και συμφωνώ με αυτούς που είπαν ε, ότι είναι πολύ σημαντική η μικροχρηματοδότηση. Το κοινωνικό ταμείο είναι γνωστό, αλλά το progress όχι και δεν έχει παρουσιαστεί αρκετά συχνά. Ωστόσο είναι βάση για όλα, για πολλά μάλλον προγράμματα και θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να προωθεί και τα προγράμματα τα οποία δεν γνωρίζουμε εξ αρχής ε, ποια θα είναι τα αποτελέσματά τους. Μπορεί δηλαδή να είναι προγράμματα που να φαίνονται λίγο επικίνδυνα στην αρχή, αλλά που τελικά ε, δίνουν ε, τεράστια αποτελέσματα. Δεν θέλουμε να σπαταλήσουμε χρήματα, αλλά να μπορέσουμε και να πειραματιστούμε. Είναι μια έκθεση λοιπόν που μας βρίσκει σύμφωνος και η Επιτροπή Έκων, στην οποία επίσης συμμετέχω, θα είχε κάθε συμφέρον να χρησιμοποιήσει την έκθεση αυτή για να υπογραμμίσει ποιες είναι οι χρήσιμες ε, δραστηριότητες της ε, ΕΤΕΠ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Δομινίκ Μαρτά. Ευχαριστώ. Ε, το είπαν οι συνάδελφοι ότι ακόμα και αν ε, ε, ε, τα, αποτελέσματα της ΕΤΕΠ είναι κάπως στο περιθώριο, ακόμα και αν τα αποτελέσματα είναι σταθερά και με το κίνδυνο να, σε, να σας εκπλήξω, Θεωρώ ότι οι προτάσεις και η έκθεση του κυρίου Κάζα είναι εξαιρετικά, άντε να μην υπερβάλλω, είναι καλές, άντε τις δεχόμαστε.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 Εξαιρετική γνωμοδότηση. Συμφωνώ με τον προηγούμενο μιλητή και θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή. Θέλω να τονίσω ένα πράγμα το οποίο πρέπει νομίζω να προσέξουμε περισσότερο. Ε, θα πρέπει ίσως να αναφερθούμε και στα δάνεια που δίνονται στους φοιτητές. Πολύ συχνά λέμε πως ε, η ευρωπαϊκή κοινωνία υποφέρει λόγω της κρίσης, αλλά όχι μόνο λόγω της κρίσης. Ε, έχουν όλοι φτωχήνη και η κινητικότητα ε, γίνεται πιο δύσκολη όλο ένα. Λέμε συχνά πως η αγορά εργασίας αναμένει ε, οι φοιτητέ να είναι πιο καλά εκπαιδευμένοι. Δεν αρκεί κανείς να είναι μηχανικός για να βρει δουλειά, πρέπει να είναι και πολύ καλός μηχανικός. Ιδιαίτερα λοιπόν στις οικογένειες όπου είναι πιο φτωχές και που δεν μπορούν ε, να χρηματοδοτήσουν την κοινωτικότητα, αυτές είναι οι οικογένειες που αξίζει να βοηθηθούν. Νομίζω λοιπόν πως θα πρέπει να είναι φιλικές ε, οι προτάσεις μας προς τους χρήστες, να ενθαρρύνουν τους νέους να πάρουν τα δάνεια αυτά και να είναι ησυχία ότι στο μέλλον θα μπορέσουν να τα ξεπληρώσουν. Ο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην παράγραφο 1, ο συντάκτη εκφράζει την ικανοποίηση ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δαπάνησε ποσό ύψου 9,1 δισεκατομμυρίων ευρώ για την προώθηση τη εκπαίδευση σε δεξιότητε και σε ευκαιρίε απασχόληση των νέων. Όμω, τι αποτελέσματα έχουν αυτέ οι πολιτικέ χρηματοδότηση. Η διάθεση των χρημάτων και ο τρόπο που χρησιμοποιούνται πόσο έχουν συμβάλει στη μείωση τη ανεργία που είναι και το ζητούμενο. Τι σημασία έχει αν έχουμε ανέργους με κατάρτιση και δεξιότητες από τους απλά ανέργους οι οποίοι δραστηριοποιούνταν σε κάποιον εργασιακό τομέα που δεν υφίστανται πια, πιστεύω ότι πρέπει να γίνει επαναξιολόγηση της πολιτικής χρηματοδότησης ούτω ώστε αυτή να συμβάλλει πραγματικά στη μείωση της ανεργίας, να δοθούν κίνητρα σε επιχειρήσεις για την απασχόληση των νέων, ούτω ώστε να σταματήσει το φαινόμενο τη εσωτερική μετανάστευση, όπου οι νέοι από τι χώρε με υψηλά ποσοστά ανεργία να αναζητούν εργασία σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Συνήθω αυτό συμβαίνει από τι χώρε του Νότου προ τι χώρε του Βορρά. Σα ευχαριστώ. Ε, thank you. Ε, Σας ευχαριστώ. Θέλει κανείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει το λόγο. Όχι. Μάλιστα, ευχαριστώ. Uh, το χρονοδιάγραμμα. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 10 Νοεμβρίου. Στην, απασχόληση, στην Επιτροπή Απασχόληση 21-22 Ιανουαρίου θα εγκρίνουμε την γνωμοδότηση και στην Ολομέλεια θα περάσει το Μάρτιο του 2015. Και τώρα να κάνουμε τις ψηφοφορίες. Έχετε τον κατάλογο, μάλλον έχετε τις κάρτες της, ε, για την ψηφοφορία. Friday will vote on the uh, European Globalization Adjustment Fund. Μάλιστα, έχουμε λοιπόν την ε, ψηφοφορία για, το... για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην κοσμιοποίηση, αίτηση ράουμα από τη Φιλανδία. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία υπέρ. Those against. Κατά. Ένας υπεραριθμός από το ΕΛΚ, παρακαλώ. Μάλιστα. Μάλιστα. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στο στρατηγικό πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασία. Και έχουμε καταρχάς ε, μία ψηφοφορία κατά τμήματα από το ΕΛΚ που την υποστηρίζει η ομάδα των φιλελευθέρων. Και μετά έχουμε ένα αίτημα για άλλη μια ψηφοφορία κατά τμήματα των φιλελευθέρων για να αφαιρεθεί η αναφορά στον ε, Αμίαντο. Εφόσον το υποστηρίζουν οι υπόλοιποι, θα την ψηφίσουμε και αυτή την, ε, το αίτημα τροπολογίας. Σε τμήματα λοιπόν, όπως είναι και στο κατάλογο ψηφοφορίας. Το σύνολο του κειμένου χωρίς την αναφορά στην έκθεση για τον αμύατο και χωρίς τις λέξεις που ζήτησε το ΕΛΚ για δεσμευτικά ευρωπαϊκά πρότυπα για το χρόνο εργασίας. Στο δεύτερο τμήμα η αναφορά στον αμίαντο, στο τρίτο κομμάτι αρχική, το αρχικό κείμενο όπως το ζήτησε το ΕΛΚ. Για το πρώτο λοιπόν, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Για το δεύτερο τμήμα, για τον αμύαντο, υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι καλά θα κάνουμε να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά αυτό. Ένα e Ένας υπεράριθμος από το ΕΛΚ. Τώρα είμαστε εντάξει και πέρας λοιπόν της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στο τρίτο τμήμα. Το δεύτερο τμήμα. As well as to develop binding work and working time. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι καλά θα κάνουμε να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Υπέρ. The vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία. Για το σχέδιο προφορικής ερώτησης. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Then we'll go to, um, Και τώρα περνάμε στο 8. Σχέδιο συμβιβασμού για την προφορική ερώτηση για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ψηφοφορία κατά τμήματα, πρώτο τμήμα. Όλο το κείμενο μέχρι το τέλος του σημείου 4. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. στο σημείο 5 του κειμένου για τις διακριτικές δράσεις. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ζητείται ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας ψηφορίας. Εγκρίνεται και περνάμε λοιπόν στην τελική ψηφοφορία. Για το σχέδιο προφορικής ερώτησης. της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στο 9. Προφορική ερώτηση λοιπόν προς το Συμβούλιο πρώτα. Υπέρ. Question to the council, access to the council? Yes. council. But here, so we here, start compromise A. Compromise A. So that's everybody okay, compromise A. Σεβασμός 8. Υπέρ. Κατά. Ε, συγγνώμη. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός B. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να αλλάξουμε ηλεκτρονικά την 7. Την τροπολογία 7. Πέρας ψηφοφορίας, λέει η Πρόεδρος. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική Συ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 11. Υπέρ κατά, άποχες, ας ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 4. Τροπολογία 12. Ε, Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα νομίζω έχει έρθει η ώρα για την τελική ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Πάλι ένας υπεραριθμός από το ΕΛΚ, σας παρακαλώ. Έχουμε λοιπόν το αποτέλεσμα πλέον. Εγκρίνεται 42 ψήφοι υπέρ. Or a question to the commission. Uh, compromise A. Who's in favour? Who's in ε, Προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή Συμβαστική A. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική B. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Άποχες απορρίπτεται. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ας ελέγξουμε παρακαλώ την ε, τροπολογία 10 στην παράγραφο 3. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική C. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα έχουμε την τελική ψηφοφορία για το θέμα αυτό. Υπέρ. Κατά αποχές. Ας κάνουμε, ας κάνουμε ηλεκτρονικά την επαλήθευση. The vote is closed. Ε, ένας υπεράριθμος από το ΕΛΚ πρωτού σας δώσουμε το τελικό αποτέλεσμα. Εγκρίνεται λοιπόν η ερώτηση αυτή. The resolution. Τώρα να ψηφίσουμε για το ψήφισμα απασχόληση και κοινωνικέ πτυχέ Στρατηγική ΕΕ για το 2020. 46. Τροπολογία 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική F. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα να περάσουμε στην τροπολογία 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 54 σε τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Έγκρινεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται να ελέγξουμε το τρίτο τμήμα. Πάλι ένα συμπεράρτημα από το ΕΛΚ. Μάλιστα. Εγκρίνεται λοιπόν. Συμβαστική G. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 61 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ, κατά, αποχές, να την ελέγξουμε, παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική H υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 64. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 65. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 66 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Με την προφορική τροπολογία. Ναι, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Δευκρίνησε η κυρία Χάρκιν. Η συμβιβαστική I, Ι, υπέρ, κατά εποχές εγκρίνεται. Και περνάμε λοιπόν στην 71. Ψηφοφορία στα τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος. Ζητείτε έλεγχος. Ένάξη ψηφοφορίας. Πέρασε. Απορρίπτεται. Καταπίπτει το δεύτερο τμήμα και περνάμε λοιπόν στην 72. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος. Έλεγχος στις 75. Έναξη ψηφοφορίας και τώρα πέρασε. Εγκρίνεται. Και περνάμε στη συμβαστική J. Υπέρ. Α, συγγνώμη, την 73 ψηφίζουμε. Την 73. Jean Lambert, 73, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στη συμβαστική J. Υπέρ. Σχόλια εκτός μικροφώνου. Yes, yes. It's, it's uh, the first uh, step. It's, it's... Στο πρώτο είναι όλο το κείμενο χωρίς τις λέξεις job quality. Υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. Στο δεύτερο κομμάτι είναι αυτές οι λέξεις. Job quality, ποιότητα απασχόλησης, υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 80. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 81. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική κάπα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 86 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Φαμ 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 87 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική L Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική. εμ, Μη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική. Α, συγγνώμη, τροπολογία 96. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 97. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται με προφορική τροπολογία για τα 6 δισεκατομμύρια, όχι εκατομμύρια. Συμβαστική νη, εν, υπέρ. Κατά. Άποχες, εγκρίνεται. Συμβιβαστική ο, όμικρον. Υπέρ. Κατά. Άποχες, εγκρίνεται. Η 109 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 110 υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 111 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Για να ελέγξουμε την 111 παρακαλώ, ηλεκτρονικός έλεγχος. Έναξη πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Α, όχι, συγγνώμη, απορρίφθηκε. 112. Πρώτο τμήμα. Κατά τμήματα, Πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 10. 113 τροπολογία. Και 114. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 115. Υπέρ. Α, καταπίπτει, καταπίπτει. αυτό. υπέρ κατά ε. αποχές εγκρίνεται 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική Q Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η ε, 125 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας κάνουμε ένα έλεγχο. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Η 126 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 127 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική R υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Εκατόν τριάντα δύο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. τριά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ας ελέγξουμε την 133 παρακαλώ, ένα ψηφορίας. Πέρας. Απορρίπτηκε. Η 134 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική S σίγμα υπέρ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 141. Με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Το αρχικό κείμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 142. Υπέρ. αποχές εγκρίνεται. 143 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 144 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 145 κατά, αποχές εγκρίνεται. 146 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος για την 146 πέρας ψηφορίας απορρίπτεται 148 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 149 υπέρ. Α, είναι συμβατή. Άρα ψηφίζουμε την 149 υπέρ. 149 υπέρ κατά απορρίπτεται. Έλεγχος ζητείται για την 149. Πέρας. Εγκρίνεται. Κατά μία ψήφο. 147 πλέον. Υπέρ. Κατά. Άποχες απορρίπτεται. 150 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 150. Ελέγχουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. 151. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. έλεγχος. Ίσως να υπάρχει διαφορετικό αποτέλεσμα. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Ήσασταν δύο τα μπροστά μου. Εγκρίνεται λοιπόν. Πολύ ωραία. Συμβιβαστική ταφ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 155 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 156 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 157 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική γιου υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 162 είναι η επόμενη υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 163 υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 164 υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 165 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 166 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 1, η τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 2, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 6. Υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται. Έλεγχο ζητείτε. Για την 6. Πέρας της 26 υπέρ. Εγκρίνεται. Η 7. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 8. Υπέρ. Έλεγχος. Η 8 λέει η πρόεδρος. Πρώτα θα ολοκληρώσουμε την ψηφοφορία για την 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ζητήσατε να ελεγχθεί η παριθμόν 7. Ο κύριος Μάρτιν. Μάλιστα, να ελέγξουμε λοιπόν την 7 ηλεκτρονικά. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρασε ψηφοφορίας. Δύο ψήφοι υπέρ. Εσείς και διπλανό σας. συγκεκριμένα. Η εννέα. Μάλλον η συμβιβαστική Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η έντεκα. υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική α, Εί. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 19 υπέρ κατά Απορρίπτεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ο κύριος Μάρτιν ζητάει το λόγο. Δεν ξέρω αν κατάλαβα. Έχω κάνει, λέει εδώ ότι έκανα μια τροπολογία γλωσσικού χαρακτήρα, αλλά εγώ απλώς συμπληρώσω το κείμενο. Την με την 21 τώρα, ναι, ναι. Αλλά απλώς ακριβώς θέλω να σας εξηγήσω. Εδώ... Α, συγγνώμη, θα την ψηφίσετε, συγγνώμη, κάνω λάθος. you have a... Νομίζω ότι έχετε παλαιό κατάλογο. Ψηφίζουμε την 21. Υπέρ για την 21 παρακαλώ. Κατά της 21. Απορρίπτεται. 22 πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε παρακαλώ. Έναξη ψηφοφορίας, πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Με τη λογική σκέψη D, 23 Μητροπολογία υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά. Άποχες Εγκρίνεται. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Φαμ 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Φεμ 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική D. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36. Υπέρ. Έλεγχος. Ρωτήτε. Την 35 θέλετε να ελέγξουμε, μάλιστα, ηλεκτρονικά. Ένταξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 36 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η ΦΕΜ 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 39. Υπέρ. Α, καταπίπτει. Καταπίπτει. Η 3... 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος. Για την 42. Έναρξη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 45. Έλεγχος για την 44. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρασε. Απορρίπτεται. Και τώρα περνάμε στη 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να ελέγξουμε και τη 45. Έναρξη. Πέρας ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Μάλιστα. Πάμε στη σελίδα 3 Τροπολογία υπαριθμών 70. Στη δική μας λίστα στην σελίδα 3, τροπολογία υπαριθμών 70.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 so we don't have to do them. They are covered. Mm-hmm. We say they are covered. Mm-hmm. Apologies for the Mm-hmm. thanks for clarifying. Mm-hmm. So we do the final vote. Mm-hmm. It Okay, it's clarified in other ways, so we don't... Μάλιστα, διευκρινίστηκε λοιπόν, δεν χρειάζεται να κάνουμε πίσω λοιπόν, να, κάνουμε, να ψηφίσουμε την 70. Τελική ψηφοφορία για το σχέδιο ψηφίσματος. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονικά να ψηφίσουμε. Have you all voted? Αν ψηφίσατε όλοι. 39 υπέρ, 5 κατά, 6 αποχές. Okay, are you ready for the next... Λοιπόν, είστε έτοιμοι για το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Πρόγραμμα ασφάλισης ε, ανέργων για την ε, Ευρώπη, το κόστος της μη Ευρώπης. Αυτή πρόκειται για μελέτη και θα δώσω το λόγο στον κύριο Τζόζεφ Ντάν, ο οποίος είναι ο Διευθυντής του Τμήματος ε, της Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας της ε, Υπηρεσίας Ερευνών, ο οποίος θα μας κάνει μια εισαγωγή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εκπροσωπώ την Υπηρεσία Ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, και τη Διεύθυνση για την Αξιολόγηση Επιπτώσεων και τις Προστιθέμενες Αξίες, η οποία συστάθηκε για να δώσει νέα εργαλεία για έλεγχο και εποπτεία στις Επιτροπές ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σήμερα λοιπόν έχουμε να σας παρουσιάσουμε μία έκθεση για το κόστος της ε, μη Ευρώπης, πηγή έμπνευσης ήταν η έκθεση του 1998 ε, του κ. Τσακίνη και ε, πλέον έχουμε και μια χαρτογράφηση του κόστους της μη Ευρώπης, όπου διαπιστώνεται ότι σε πολλούς τομείς επιπλέον δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορούσαν ίσως να αποτελέσουν όφελος για την Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα τις τάξεις του 1-3 ε, ευρώ. Και θεωρούμε ότι ένα τμήμα αυτών θα μπορούσε να προκύψει από πρωτοβουλίες όπως ε, το κοινό σύστημα ασφάλισης για τους ανέργους. Δεν κάνουμε κάποια συγκεκριμένη σύσταση, αλλά ε, στόχος μας είναι να σας βοηθήσουμε και να σας δώσουμε τα απαραίτητα εργαλεία προκειμένου να υπάρχουν αυτές οι αναλεκτικές λύσεις ως προτάσεις. Ε, είχαμε το Φεβράριο του 2014 το σχέδιο της μελέτης, έγινε μια σύντομη συζήτηση τίποτε. Τότε και έκτοτε θεωρώ ότι έχει αυξηθεί η σημασία του θέματος. Ε, υπάρχουν αρκετές ε, ε, συζητήσεις σε πολιτικό επίπεδο αλλά και οικονομικές εξελίξεις που το καταδεικνύουν αυτό. Έχουμε δύο παραρτήματα. Το ένα το έχει ετοιμάσει η ΣΕΠΣ και έχει κάνει μια προσωμείωση και το δεύτερο το Κέντρο Οικονομικής Έρευνας στο Μόναχο και προτείνουμε να ακούσουμε τις δύο παρουσιάσεις. Ο καθής από τους εμπειρογνώμονες θα μιλήσει για 7 λεπτά και θα ήθελα να σας πω εν παρόδο ότι ίσως και ε, στην έκθεση να αναφερθούμε στην εμπειρία των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία έχει κάποιο ενδιαφέρον στο πλαίσιο αυτό, δεδομένου ότι υπάρχει ένα σύστημα ασφάλισης ανέργων ε, σε λειτουργία και ε, ήρθαμε σε επαφή και με το, ε, το Γραφείο Προπολογισμού και το Γραφείο Ερευνών του Κογκρέσου που ασχολούνται με τα θέματα αυτά και αυτό είναι ένα από τις σημαντικές εναλλακτικέ λύσεις ε, εάν θέλουμε πραγματικά να υλοποιήσουμε αυτό το στόχο. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα ακούσουμε τους δύο πυρογνώμονες και ε, θα δείτε παρουσιάσει σε PowerPoint. Ωραία. Ο κύριος Τζόνς θα μας κάνει την παρουσίαση. Παρακαλώ. Um, actually, I'm Ilaria Masai, I live εγώ είμαι η Λάρια Μασέλη από το ΣΕΠΣ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την πρόσκληση και για το γεγονός ότι μας ε, αφήνετε να σας παρουσιάσουμε τη μελέτη μας ε, για την ε, ασφάλιση των ανέργων, που θεωρούμε ότι πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για τον Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταρχάς να ξεκινήσουμε από το βασικό ερώτημα. Ασφάλιση για ποιο λόγο. Υπάρχει συνεχής βιβλιογραφία, αυξάνεται συνεχώς και έχουμε προτάσεις για δύο σκοπούς. Ένα κατά της λεγόμενης ε, βροχής των Βρυξελών που θα ε, φέρει ένα περιορισμένο ένα περιορισμένη έκτασης ε, σοκ. Το ταμείο αυτό θα παρεμβαίνει λοιπόν για ε, επιδόματα ανεργίας για περιορισμένο χρονικό διάστημα στις ε, χώρες που πλήττονται από την ανεργία για τους ε, ανέργους. Και υπάρχει και ένα δεύτερο στοιχείο που διαπιστώσαμε στο ΣΕΠΣ, διαπιστώσαμε ότι προκειμένου να καλύψουμε τα μεγάλα σοκ, δηλαδή αν αφήσουμε τα συνηθισμένα στο εθνικό σύστημα ασφάλισης και δημιουργήσουμε ένα ταμείο το οποίο ουσιαστικά είναι μια δεύτερη ασφάλιση ε, για κάλυψη σε περίπτωση που έχουμε έναν ε, ανεμοστρόβιλο φαινομένων. Η βασική υπόθεση είναι ότι θεωρούμε ότι το κόστος της ύφεσης με αύξηση της ανεργίας κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες είναι πάνω από το διπλάσιο της ύφεσης αν έχουμε ανεργία ε, αυξανόμενη κατά δύο μόνο ποσοστιαίες μονάδες. Και πώς λειτουργεί αυτό. Έχουμε ένα τύπο, όπως βλέπετε εδώ στη διαφάνεια. Είναι πολύ απλός ο τύπος. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο παρεμβαίνει για να χρηματοδοτήσει τα επιδόματα ανεργίας σε μια χώρα όταν το ποσοστό της ανεργίας αυξάνεται άνω ενός συγκεκριμένου ορίου. Και εδώ ο τύπος μας λέει ότι θεωρούμε ότι το Ταμείο θα πρέπει να πληρώνει επιδόματα ανεργίας για τους ανθρώπους που μένουν για μικρό διάστημα άνεργοι όταν το ποσοστό αυτών των ανέργων πηγαίνει πάνω από κάποιο όριο. Και ουσιαστικά αυτό είναι το ποσοστό των ε, μακρόχρονων ανέργων ε, συν ένα ποσοστό. Αυτό το συν μπορεί να είναι διαφόρων περιπτώσεων. Έχουμε διάφορες περιπτώσεις που μπορείτε να ε, έχουμε, βλέπετε εδώ, αν είχαμε αυτό το φαινόμενο από το 2000. Ουσιαστικά λοιπόν ένα ταμείο για να αντιμετωπίσει ένα σοκ τύπου βροχή των Βρυξελών θα σημαίνει ότι έχουμε 161 ε, διαφορετικές περιπτώσεις που θα μπορούσαν να είχαν συμβεί στα προηγούμενα 12 χρόνια. Και αυτό προκύπτει ως ένευσμα ε, μιας ε, σύντομης περίοδου ανεργίας και μας οδηγεί σε μια απόκληση της τάξης του 0,1. Ε, όταν έχουμε ε, πάνω από 4% ανεργία, σε αυτή την περίπτωση το Ταμείο θα παρέμβει 90 φορές σε 12 χρόνια και μετά έχουμε πλέον ε, τον ανεμοστρόβιλο όπως τον αποκαλούμε και σε αυτή την περίπτωση οι παρεμβάσεις από το Ευρωπαϊκό Ταμείο είναι πιο σπάνιες μεν αλλά πιο σημαντικές και αυτό θα συνέβαινε σε 40 περιπτώσεις. Έχω εδώ δύο διαγράμματα για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχουμε την Ελλάδα και την Εστονία. Ε, προφανώς και το Ταμείο θα είχε παρέμβει στην Ελλάδα στη διάρκεια της μεγάλης ύφεσης και θα είχε βοηθήσει τη χώρα με συνεισφορά της τάξης του 1% ε, του ΑΕΠ κάθε χρόνο. Σχεδόν 1% κάθε χρόνο. Η περίπτωση της Εστονίας είναι ενδιαφέρουσα διότι μα δείχνει ότι η μεγάλη ύφεση δεν ήταν μόνο η μόνη ενδιαφέρουσα περίπτωση. Στην περίπτωση της εμφαν... Ε, Εστονίας δεν θα είχε παρέμβει μόνο το 2009 και το 2010 ή το 2002 και το 2003 που είχαμε ε, και πάλι προβλήματα στη χώρα. Να σας πω ποια είναι τα απλεονεκτήματα αυτού του Ταμείου ε, Πρόσθετης Ασφάλισης. Καταρχά, θεωρούμε ότι είναι εφικτό από πολιτική σκοπιά. Είναι πολύ εύκολο να το δημιουργήσουμε αντί να έχουμε ένα τεράστιο ε, πρόγραμμα επιδομάτων ανεργία πανευρωπαϊκά. Και ο λόγο είναι ότι ε, δεν θα χρειάζεται πολύ χρηματοδότηση. Η εκτίμησή μα είναι ότι το μεγαλύτερο ποσό του Ταμείου θα ήταν για το 2009 όπου είχαμε πολύ σοβαρές περιπτώσεις και εκεί θα χρειαζόμασταν 30 δισεκατομμύρια που είναι περίπου 0,3% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Με αυτή την σχετικά μικρή συνεισφορά λοιπόν θα είχαμε πολύ σημαντικές συνέπειες ε, στις χώρες που αντιμετώπιζαν κρίση. Αλλά επίσης θα ήταν και εύκολη διαχείριση γιατί ουσιαστικά θα λειτουργούσε αυτόματα. Κάθε φορά που υπερβαίνει το ποσοστό της ανεργίας σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο μπορεί να υπάρξει παρέμβαση με σχετικά λίγη γραφειοκρατία. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι αυτή τη μορφή στο ταμείο θα μπορούσε ίσως να συμβαδίζει και με τη σύγκληση ε, του εθνικού συστήματος, διότι όπως έχει καταδείξει η έρευνα των συναδέλφων εδώ, ε, δεν λειτουργούν όλα τα προγράμματα επιδομάτων ανεργίας με τον ίδιο τρόπο. Σε κάποιες χώρε χώρες βοηθούν στη σταθεροποίηση της οικονομίας και σε κάποιες άλλες ε, λιγότερο. Και φυσικά υπάρχουν και προσκόμματα. Ένα πρόσκομα είναι το γεγονός ότι το Ταμείο θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αποφασιστεί ότι καλύπτει την Ευρωζώνη ή την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, ε, όποια ομάδα και να αποφασιστεί, εκ των δύο θα πρέπει να υποχρεωτική συμμετοχή. Και ο λόγος είναι συγκεκριμένος. Αν ε, δεν είναι υποχρεωτική η πρόσθετη ασφάλιση, τότε μόνο ε, οι κακοί ε, εντός εισαγωγικών θα ε, θέλουν να συμμετέχουν στο Ταμείο. Ένα άλλο πρόσκομα το οποίο προέκυψε αρκετές φορές στη διάρκεια των μελετών μας είναι ο φόβος των μόνιμων επιδομάτων. Εμείς θεωρούμε ότι αυτός ο φόβος δεν είναι αιτιολογημένος διότι αν δούμε ένα διάστημα αρκετά μεγάλο ώστε να έχουμε αποτελέσματα, θα δούμε ότι αργά ή γρήγορα ε, κάθε χώρα αντιμετωπίζει μεγάλα σοκ από πλευρά ανεργία. Παραδείγματο χάρη, αν το είχαμε από τη δεκαετία του 90 το σύστημα, οι χώρε ε, που θα είχαν υποφαληθεί τότε θα ήταν η Δανία και η Σουηδία, που κανεί δεν διανοείται σήμερα ότι θα ήταν χώρε κρίση, αλλά τότε αντιμετώπισαν ένα πολύ σοβαρό ε, πρόβλημα στι αρχέ τη δεκαετία του 90 και θα του είχε βοηθήσει το Ταμείο αν υπήρχε. Δύο λόγια τώρα για να φερθώ στο σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών που εμείς θεωρούμε ότι δεν μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για την Ευρώπη. Και ο λόγος είναι ότι τα προγράμματα ασφάλισης ανέργων ε, στις Ηνωμένε Πολιτείε έφτασαν σε ομοσπανδιακό επίπεδο διότι υπήρχε φόβος κοινωνικού ντάμπινγκ μεταξύ των διαφόρων πολιτιών. Ε, ο φόβος αυτός είναι πολύ μικρότερος ε, διότι... Ε, ούτως ή άλλως ε, είχαμε ασφάλεια για τους ανέργους ε, ε, εδώ και αρκετά χρόνια στην Ευρώπη και αναπτύχθηκε παρά τους φόβους που υπήρχαν για αυτά τα προβλήματα. Ο άλλος λόγος είναι ότι το σύστημα ανεργίας στις ΗΠΑ έχει και ένα προπολογισμό ευελιξίας για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Δηλαδή, αν θεωρήσουν ότι χρειάζεται, μπορούν να επεκτείνουν τους πόρους. Και εμείς δεν θεωρούμε ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να αντιδράσουν τόσο γρήγορα σε περίπτωση ύφεσης. Παρόλα αυτά, Μία ε, σύστασή μας ε, έχει εμπνευστεί από το σύστημα των ΗΠΑ και είναι ε, το λεγόμενο experience rating κάθε πολιτεία στο σύστημα των ΗΠΑ συνεισφέρει στο Ομοσπονδιακό αυτό ταμείο. Και σε περίπτωση που υπάρχει κρίση μπορούν να δανειστούν από αυτό το μεγαλύτερο ταμείο υπό την προπόθεση ότι θα επιστρέψουν τα χρήματα. Επομένω υπάρχει μια εξισορρόπηση του οικονομικού κύκλου και ακριβώ ε, και εμεί θεωρούμε ότι για να μην έχουμε μόνιμε μεταφορέ θα πρέπει να υπάρχει ο συγκεκριμένο κανόνα. Μια τελευταία παρατήρηση ο συνδυασμός του προγράμματος αυτού με άλλα προγράμματα. Αυτό που μας δείχνει η έρευνα είναι ότι τα επιδόματα ενεργείας σχεδιασμένα με κάποιο τρόπο είναι πολύ καλά μεν, αλλά ε, είναι πολύ πιο αποτελεσματικά όταν συνδυαστούν και με άλλα προγράμματα. Τα κονδύλια λοιπόν του Ευρωπαϊκού Ταμείου για επιδόματα ενεργείας θα πρέπει να συνδυαστούν και Ε, με μία ε, σειρά από προγράμματα για τα ε, Ιδρύματα της Αγοράς Εργασίας. Ευχαριστώ κυρία Μασίλη. ο κύριος Τζόουνς. Uh, Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ που μας καλέσατε στην γραμματεία. Ονομάζομαι Νόιμαν και να σας πω ότι τα όσα θα σας παρουσιάσω προέρχονται από ευρωπαϊκές έρευνες.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 Εδώ έχουμε μια συγκεκριμένη περίοδο προσωμείωσης αλλά και διάφορες εναλλακτικέ που, στις οποίες έχουμε καταλήξει με τη βοήθεια των ασφαλιστικών συστημάτων. Πριν σας μιλήσω για την προσωμείωση που κάνουμε θα ήθελα να σας παρουσιάσω το γενικό σχεδιασμό ε, των επιλογών που έχουμε όσον αφορά τη, τα ταμεία ενεργείας στην περιοχή μάλλον της Ένωσης βασική ασφάλιση λοιπόν έχουμε ένα μήνυμο επίπεδο ασφάλισης εγγυημένο. Για το δεύτερο σύστημα, το συμπληρωματικό σε εθνικό επίπεδο, μιλάμε για, πιο, για περισσότερα επιδόματα που αυξάνουν τις, την, τις επιδράσεις της ασφάλισης για μακρές περιόδους ύφεσης. Μπορούμε να σκεφτούμε δε όσον αφορά τη χρηματοδότηση για ένα σύστημα με ή άνευ βαθμολόγηση της προηγούμενη εμπειρία ή μπορούμε να μιλήσουμε για μηχανισμούς ανάκλησης. Όσον αφορά τα επιδόματα, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε τα διαρκή ή τα αυτά που ξεκινούν με, ε, συγκεκριμένο αίτιο για το δεύτερο αυτό σκέλος μιλάμε για συγκεκριμένα επιδόματα τα οποία ε, ξεκινούν όταν πρόκειται για σημαντική οικονομική κρίση. Έχουμε δηλαδή τρεις βασικές επιλογές. Μια βασική ε, ασφάλιση ανεργίας, επιδόματα ανεργίας αλλά και ε, πλέον επιδόματα τα οποία δίνονται εάν και εφόσον ισχύουν κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Για τη βασική, λοιπόν, το βασικό σύστημα ανεργίας, επιδομάτων ανεργίας, αυτό είναι ε, αυτό που καλύπτει αποκλειστικά και μόνο την ανεργία. Ε, μειώνεται σε μακρές περιόδους ύφεση. Όμως τα επιπλέον επιδόματα ξεκινούν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα και εξασφαλίζουν σε περίπτωση ε, μεγάλων περιόδων ύφεση. Τα δε επιπλέον επιδόματα αυτά ξεκινούν ε, πάνω από κάποιο ε, κατόφλι. Δεν υπάρχει κάποιος μόνιμος τρόπος κατανομής τους, ακριβώς επειδή στόχο έχουν συγκεκριμένους τύπους ανεργίας. Θέλω να είμαι σύντομο, γι' αυτό περνώ στο επόμενο, επόμενο ε, διαφάνεια. Αν δούμε τώρα τα θέματα κινδύνου, εδώ έχουμε τις, ε, τα, συστήματα ασφάλισης που καλύπτουν ε, τα επιδόματα ενεργείας. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο οι εθνικές κυβερνήσεις εξακολουθούν να μπορούν να φέρουν το βάρος της καταβολής αυτών των αποζημιώσεων. Μετά πρέπει να δούμε αν τα επιδόματα ενεργείας θα πρέπει να βγουν από το κοινό κορβανά ε, και έπειτα θα πρέπει να δούμε και θέματα διοικητικής χειραγώγησης, αλλά όπως σας είπα θέλω να είμαι ε, σύντομος. Για το βασικό σύστημα κάλυψης επιδομάτων ανεργίας ε, θα πρέπει να δούμε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, το οποίο συζητάται σε πολιτικό αλλά και σε ακαδημαϊκό περιβάλλον. Αυτό που κάνουμε στην ανάλυση μας ε, διερωτώμεθα εάν υπήρχε ένα τέτοιο βασικό σύστημα για την κάλυψη των επιδομάτων ανεργίας από το 1999 και υπολογίζουμε ε, τι θα γινόταν από το 2000 μέχρι το 2013. Προσωμιώνουμε λοιπόν όσον αφορά την κάλυψη, υπολογίζουμε ότι 50% των μεικτών εισοδημάτων αντικαθίσταται ή ε, μάλλον είναι εγγυημένα από το σύστημα ασφάλισης και έτσι αυτό θα ε, γινόταν σε επίπεδο χωρών και όχι σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα υπήρξε καταβολή, υπήρχε καταβολή ενός ε, φόρου επί των εισοδημάτων κατά 1,6% για κάθε εισόδημα από απασχόληση. Θα είχαμε λοιπόν ε, ε, θα είχαμε 49 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο Εξετάζουμε τα εναλλακτικά σενάρια όσον αφορά την βαθμολόγηση, την εμπειρία, στη ρήτρα ανάκληση, μάλλον, μάλλον ε, εκ των υστέρων προσαρμογών στις ε, φορολογικές ε, ε, Και τώρα θα δώσω το λόγο στον Ματίας Ντόλς. Σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ που προσπαθείτε να περιορίσετε το χρόνο σας για τις παρεμβάσεις σας. Όμως οι μεταφραστές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να σας παρακολουθήσουν. Οπότε αν μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο αργά. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα συνεχίσω παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της προσωμείωσης της ανάλυσής μας και θα ξεκινήσω με το ποσοστό κάλυψης που βασικά είναι, αφορά την ΟΝΕ ναι και το τι επιρροή θα είχε το δικό μας σχέδιο. Με τη μπλε γραμμή βλέπουμε την εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία και Γερμανία. Οι τέσσερις αυτές χώρες, ε, κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, είναι παραδείγματα όπου υπήρχαν αποκλίνουσες τάσεις στην απασχόληση σε αυτή τη χρονική περίοδο. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, το ποσοστό ανεργίας αυξανόταν μέχρι το 2005 και τότε ήταν το δεύτερο ψηλότερο στην Ευρωζώνη, ενώ το ποσοστό ανεργίας ήταν σχετικά χαμηλό σε άλλα κράτη-μέλη. Και έπειτα, ξεκινώντας με την ελληνική ύφεση, η, ε, τα ποσοστά ανεργίες αυξήθηκαν κατακόρυφα στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιλλανδία, ενώ σχεδόν σταθερά μειώνονταν στην Γερμανία. Αυτό που βλέπουμε με την κάλυψη, με την πορτοκαλί γραμμή, είναι ότι ένα πρόγραμμα από το οποίο θα κάλυπτε τα επιδόματα ενέργειας θα έπρεπε να καλύπτει ε, και μακρές περιόδους ύφεσης λόγω του μεγάλου μεριδίου μη επιλέξιμων ε, μακροχρόνιων ανέργων. Συνεχίζουμε με τις επιπτώσεις ε, στη δημοσιονομικά και τις, και τις ροές. Σε αυτό το γράφημα βλέπουμε μέση ετήσια καθαρή συνεισφορά για τα ίδια αυτά χρόνια και στις περισσότερες χώρες μέλη θα είχαν ε, θα, συνέβαλαν καθαρά σε, για κάποια χρόνια ενώ θα, θα ε, δέχονταν καθαρά χρήματα σε κάποιες άλλες χρονιές. Η Γερμανία, για παράδειγμα, το 2004 και 2005. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη που μονίμως θα συνέφεραν. Και αυτό ισχύει για την Αυστρία και την Ολλανδία ή που θα ήταν αποδέκτες ε, μονίμως, όπως η Γαλλία, η, Λα... Λετωνία και η Ισπανία. Θα πρέπει ωστόσο να λάβουμε υπόψη ότι έχουμε λάβει υπόψη μια περίοδο προσωμείωσης 13... 13 χρονών και τα αποτελέσματα θα μπορεί να ήταν και διαφορετικά αν είχαμε πιο μακροχρόνια περίοδο. Τώρα, αν υπήρχε αυτόματο σταθεροποίηση σε κεντρικό επίπεδο, σταθεροποιητή, διαπιστώσαμε ότι αυτό το πρόγραμμα θα είχε απορροφήσει ένα μεγάλο κομμάτι του σοκ του 2009. 46% των μέτρων αυτών ε, της μείωσης των εισοδημάτων θα είχε απορροφηθεί σε επίπεδο ευρωζώνης και επίσης σε αυτό το γράφημα βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη τα οποία χτυπήθηκαν περισσότερο στη διάρκεια της κρίσης, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία, ένα μεγάλο τμήμα του σόκου θα είχε απορροφηθεί στις αρχές της κρίσης, αν και όπως συνάδελφε και ο συνάδελφος Νόημαν λόγω της κυκλικής ανεργίας αυτό το εφέ σταθεροποίησης θα είχε μειωθεί τις επόμενες χρονιές λόγω της αύξησης των μακροχρόνια άνεργων. Επίσης λάβαμε υπόψη διάφορες άλλες μεταβλητές αυτής της βασικής, ε, του βασικού προγράμματος ε, για την ΟΝΕ. Ένα πρόγραμμα δηλαδή όπου τα επιδόματα διατηρούνται στο διατηρούνται στο 50% των ε, μισθών. Στην ουσία θα πρέπει να δούμε δηλαδή τι θέλουμε καλύτερα, αυτόματη σταθεροποίηση και, ή αυτόματη ανακατανομή. Δηλαδή όσο λιγότερο γενναιόδωρο είναι το πρόγραμμα, τόσο λιγότερη σταθεροποίηση παρέχει. Να προχωρήσω στην αξιολόγηση της εμπειρίας και τον μηχανισμό ε, εκ των προσαρμογής. Αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ είναι πώς θα είχαν οι συμβολές, οι εισφορές μάλλον, αν αυτές βασίζονταν σε τρεις διαφορετικές ε, ε, ε, περιστάσεις. Δηλαδή, αν είχαμε καθαρό, καθαρή εισφορή, την μπλε γραμμή όπου έχουμε ομοιόμορφη συμβολή σε επίπεδο ευρωζώνης και εκεί που έχουμε διαφορετικούς μηχανισμούς με συγκεκριμένους ε, συγκεκριμένη σταθερή ε, εισφορές. Μπορούμε λοιπόν να δούμε ότι η αυτόματες προσαρμογές και ο μηχανισμός εκ των υστέρων προσαρμογής θα περιόριζε τις ε, διασυνοριακές ε, συναλλαγές. We consider um, schemes, contingent benefit schemes, which are... Τέλος, βλέπουμε συγκεκριμένα προγράμματα για επιπλέον επιδόματα αν η ενεργεία αυξηθεί κατά 1% στον πρώτο χρόνο, εδώ έχουμε την, πράσινη γραμμή, ή αν αυξηθεί στα δύο τελευταία χρόνια, δεύτερη πιθανότητα, ή αν αυξηθεί η ανεργία κατά 1% τα τελευταία τρία χρόνια. Έχουμε διάφορα δηλαδή προγράμματα με διάφορες ε, ε, ε, περιόδους ιστορικής αναδρομής. Αυτό που προέκυψε από αυτή την ανάλυση είναι ότι και το επίπεδο των διασυνοριακών μεταφορών θα περιοριστεί με αυτά τα προγράμματα που προβλέπουν συγκεκριμένες στοχοθετημένες μεταφορές για τις χώρες που έχουν χτυπηθεί από την αυξανόμενη ενεργεία. Να τονίσω για παράδειγμα πως η Γαλλία που είναι αποδέκτης στην δική μας προσωμείωση θα μετατρεπόταν σε ε, καθαρό ε, ε, δότη. και η Ισπανία θα ήταν καθαρός δότης ανάμεσα στο 2000, μέχρι το 2007 ή καθαρός αποδέκτης μόνο από το 2008 και ύστερα. Συμπέρασμα είναι ότι μια ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα επιδομάτων ανεργίας θα ενίσχυε και τον προπολογισμό αλλά και την κοινωνική διάσταση της ευρωπαϊκής πολιτικής. Θα μπορούσε αυτό να σημάνει μια αναλλαγή, αυτό θα μπορούσε να εφαρμοστεί με σχετικά μικρό κόστος ενώ θα είχε μεγάλα κέρδη, 49 δις ετησίως και βέβαια εξαρτώνται όλα αυτά από τις τάσεις της ανεργίας στα διάφορα κράτη-μέλη. Ε, Και τέλος, όπως ήδη είπα, η ε, αυτόματη σταθεροποίηση θα αυξανόταν πολύ με βάση αυτά τα προγράμματα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ε, Εγώ ευχαριστώ πολύ. Τη μελέτη αυτή την κάνατε κατόπιν ετήματος της Επιτροπής Απασχόλησης και δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας για συζήτηση. Αλλά τέλος πάντων θα ήθελα να δώσω το λόγο σε όσους ενδιαφέρονται. Αν θέλουν να σας θέσουν ερωτήσεις ή να κάνουν παρατηρήσεις. Θα ξεκινήσω. Από τον κύριο Μπέκερ, από το ΕΛΚ, θέλετε το λόγο. Όχι, τότε για το ΣΤΕΜ. Καταρχάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ε, πληροφορίες ε, από το 2008 το θέμα αυτό της ασφάλισης των ανέργων πλανάται έτσι γενικά στην Ευρώπη και εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει η όρος ασφάλιση των ανέργων γιατί στη Γερμανία προκαλεί αντανακλαστικά απόρριψη. Σκεφτόμαστε πιο πολύ ε, μηχανισμούς αλληλεγγύης Νομίζω ότι θέσατε βασικά θέματα τα οποία είναι σημαντικά και για μας. Είπατε ότι υπάρχουν ε, κάποιες πλούσιες χώρες οι οποίες ε, το 2005 στο 2008 ήταν αυτοί που κέρδισαν από την ασφάλιση των ενέργων. Ε, κοίταξα τα αριθμητικά στοιχεία στη Γερμανία και διάφορες λοιπόν μελέτες δείχνουν ότι η, Γερμανία είχε τους πόρους σε δύσκολους καιρούς για θέματα ασφάλισης και των ενέργων. Για μας αυτό που είναι σημαντικό είναι το εξής. Μέσω μιας ευρωπαϊκής ρυθμίσης για την ε, ασφάλιση των ενέργων μέσω ενός ε, μηχανισμού αλληλεγγύης, να φροντίσουμε να μην υπάρχει αρνητικό κόστος για τους εργαζόμενους. Παρόλα αυτά υπάρχει, υπάρχει και η πιθανότητα να καταλήξουμε σε ελάχιστα πρότυπα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό είναι κάτι το ευκταίο. Ρωτώ λοιπόν από δική μου πλευρά, πιστεύετε ότι υπάρχουν θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις σε ό,τι αφορά την κατανομή των ε, εισοδημάτων στα κράτη-μέλη. Και αληθεύει αυτή η εκτίμηση ότι μέσω της ασφάλισης των ανέργων σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα καταλήγαμε σε ένα ευρωπαϊκό σύστημα ελάχιστων προτύπων, κάτι που είναι εξαιρετικά ευκταίο. Ύστερα, υπάρχουν διάφοροι επικριτές της Ευρώπης που ε, υπογραμμίζουν τις καταχρήσεις. Πώς μπορούμε λοιπόν εκ των προτέρων να αποκλείσουμε τέτοια ενδεχόμενο καταχρήσεων. Ε, we'll take second question and Ακούσουμε και μια δεύτερη ερώτηση και μετά θα απαντήσετε. η κυρία Χάρκιν, εκ μέρους των Φιλελευθέρων. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και τους ομιλητές. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Αποτελούν σίγουρα τροφή για σκέψη και πάντα είναι χρήσιμο να υπάρχουν προσωμιώσεις οι οποίες μας επιτρέπουν να έχουμε μια εικόνα για τις συνέπειες, διότι ορισμένες φορές έχουμε πολύ ωραίες ιδέες ή θεωρούμε ότι είναι πολύ ωραίες οι ιδέες μας και μετά τις ελέγχουμε και διαπιστώνουμε ότι οι συνέπειες δεν είναι πάντα τόσο θετικές όσο είχαμε θεωρήσει. Ορισμένες φορές είναι και εντελώς το αντίθετο αυτό που περιμέναμε. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Θεωρώ ότι είναι χρήσιμο που γίνεται αυτή η συζήτηση. Τώρα, επειδή εγώ βλέπω το όλο θέμα από ένα πρίσμα πολύ περιορισμένων γνώσεων επί του ζητήματος. Έχω κάποιες ερωτήσεις λοιπόν, τις οποίες θα ήθελα ε, να σας θέσω. Υπάρχει εξή παρατήρηση. Αναφερθήκατε στο σκεπτικό της μόνιμης ε, μεταφοράς αυτών των επιδομάτων. Νομίζω ότι η πρώτη ομιλήτρια που αναφέρθηκε ε, σε αυτό, αν είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, δεν υπάρχει μόνιμη μεταφορά ή τουλάχιστον είναι ελάχιστη η δυνατότητα ελαχιστη μόνιμη μεταφορά. Ε, πρέπει να το εξετάσω, αλλά είναι πολύ σημαντική αυτή η παρατήρηση. Ε, ο τελευταίος ομιλητής, κοιτάζω εδώ και τα συμπεράσματα τη παρουσίασή σας, Αναφερθήκατε σε, αναφέρθηκε σε μηχανισμούς ε, ε, εκ των υστέρων αλλαγής. Φαντάζομαι ότι άμα το διαβάσω θα καταλάβω τι εννοεί, αλλά ε, θα μπορούσατε να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω εσείς. Τι συνέπειες θα έχει αυτός ο μηχανισμός. Έχω πάρα πολλές άλλες ερωτήσεις, αλλά αυτή τη στιγμή τώρα τα διαβάζω και ίσως θα μπορούσα να επανέλθω αργότερα με το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ και πάλι για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Ο κύριος Μάν. Είναι θετικό το γεγονό ότι το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη τι κοστίζει το να μην υπάρχει η Ευρώπη γιατί νομίζω ότι μας ε, διακρίνει εμάς που είμαστε εδώ και καιρό στην, ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από αυτούς που μόλις έχουν έρθει και μας λένε ότι ας την καταργήσουμε την Ευρώπη. Δυστυχώς ε, αυτή η άποψη είναι πολύ δημοφιλή σε κάποια κρατημέλη. Μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό και θα το αλλάξουμε πιστεύω αν ε, είμαστε επιτυχεί. Συμφωνώ με την ιδέα του Γιούγκερ ότι χρειαζόμαστε καινούργια μέσα, χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, αλλά σε θέματα εφαρμοσιμότητας. Και αυτό που θέλω να το πω σε όλους τους εμπειρογνώμονες, για να υπάρχει αυτή η ευρωπαϊκή ασφάλιση, θα πρέπει να αλλάξουν τα εθνικά συστήματα ασφάλισης. Είμαστε πρόθυμοι να το κάνουμε αυτό. Και θα πρέπει να λάβουν διαφορετική διαμόρφωση οι εθνικές, ε, τα εθνικά συστήματα. Δεν υπάρχει ενιαία ε, ευρωπαϊκή αγορά. Υπάρχουν και κοινωνικοί εταίροι οι οποίοι δεν διαπραγματεύονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και απλά δίνουν την εμπειρία του κάθε κράτους μέλους. Δεν υπάρχει λοιπόν ο κίνδυνος να υπάρξει μια νέα ένωση μεταφορές, γιατί έχει δίκιο η Γιούτα Στάινρουκ. Πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη, αλλά έχουμε και μέσα, έχουμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ύψους εκατομμυρίων, εκατομμυρίων Έχουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Έχουμε επαρκή μέσα που ήδη υφίστανται. Δεν διατρέχουμε τον κίνδυνο να είμαστε υπεύθυνοι για τους ανέργους άλλων χωρών. Αυτό δεν μπορεί να είναι το επισημητό. Ναι, λοιπόν, να ενισχύσουμε την κοινωνική διάσταση, αλλά να μην υπάρξει ένα μεγάλο σύστημα χρηματοδότησης, γιατί θα δημιουργήσουμε λανθασμένες προσδοκίες. Να πούμε απλά ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τα συστήματα που ήδη υφίστανται. Έχουμε επαρκή ευρωπαϊκά μέσα, τα οποία ήδη λειτουργούν. Έχω μεγάλες αμφιβολίες. Αν θα μπορούσατε λοιπόν να ε, απαντήσετε σε αυτά τα θέματα που με απασχολούν. Ευχαριστώ πολύ. Αν θα θέλετε να ξεκινήσετε και να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ για την παρατηρήση και για τις ερωτήσεις αυτές. Να ξεκινήσω από το τέλος, από την τελευταία παρουσίαση. Συμφωνώ απόλυτα ότι όταν ε, μιλάμε και σκεφτόμαστε θέματα εφαρμογής και το πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί μια ευρωπαϊκή ασφάλιση, με ποιους όρους. Όντως, ε, ο δρόμος είναι πάρα πολύ μακρύς. Και σίγουρα θα σήμαινε εναρμόνιση των υφιστάμενων θεσμών στον τομέα της αγοράς εργασίας. Σίγουρα δηλαδή δεν είναι ένα μέσο το οποίο μπορεί να εισαχθεί βραχυπρόθεσμα. Αυτό που θα ήθελα ωστόσο να επισημάνω είναι το εξή. Τα εφιστάμενα μέσα τα, υπάρχουν, τα οποία υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχουν αυτόματη λειτουργία σταθεροποίηση και αυτή είναι η ιδέα λοιπόν μιας ευρωπαϊκής ασφάλισης ε, να υπάρχει ένας μηχανισμός σταθεροποίησης και οι μηχανισμοί αυτοί να έχουν και μια συνιστόσα οικονομικής σταθεροποίησης. Ένα τέτοιο μέσος λοιπόν αυτόματης σταθεροποίησης δεν υπάρχει σε επίπεδο Ευρωζώνης ως σήμερα και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση είναι μη τυπική ένωση γιατί σε άλλες τέτοιες νομισματικές ενώσεις υπάρχουν κεντρικά τέτοια μέσα ενώ στην Ευρωζώνη δεν υπάρχει. Παρ' όλα αυτά Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος της ηθικού ρίσκου, των, ε, της μόνιμης μεταφοράς χρημάτων. Είναι, θέματα υφιστάμενα αυτά και τα οποία θα πρέπει να οργανωθούν ε, άλλωστε και να συζητηθούν. Ύστερα, μου ζητήσατε να σας εξηγήσω το μηχανισμό που βασίζεται στο experience rating. πληρωμές ή ε, συνεισφορές για την ασφάλιση των ε, ανέργων δεν ταυτίζονται σε ό,τι αφορά το ποσοστό τους, το συντελεστή τους σε όλα τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν κράτη-μέλη που είναι μεγάλες μεταφορές και που προσαρμόζεται ο συντελεστής στον οικονομικό κύκλο για να υπάρξει ουδετερότητα σε επίπεδο κρατών μελών. Ένας μηχανισμός ο οποίος θα μπορούσε να οδηγήσει στον περιορισμό του κύκλου μεταφορών μεταξύ κρατών μελών. Για την πρώτη παρέμβαση να κάνω κάποια σχόλια. Σε ό,τι αφορά την, τον αντίκτυπο στην κατανομή. Αυτό είναι λίγο δύσκολο να το προσωπικοποιήσουμε όσο υπάρχουν εθνικά μέλη. Αυτή η, ιδέα της ε, βασικής ασφάλισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να αντικαταστήσει εν μέρη τα εθνικά συστήματα ασφάλισης. Εδώ είναι δύσκολο να κάνουμε εκτιμήσεις, γιατί θα πρέπει να κοιτάξουμε πρώτα πώς διαμορφώνονται τα εθνικά συστήματα. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις. Σε ό,τι αφορά την δυνατότητα και το ενδεχόμενο καταχρήσεων, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή ότι στην περίπτωση αυτή σίγουρα θα χρειάζεται εναρμόνιση των ε, σχετικών θεσμικών αρχών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εφόσον επιθυμούμε να υπάρχει τέτοιο σύστημα ευρωπαϊκής ασφάλισης ανέργων. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. Αν δεν τις απαντήσουμε όλες, να μας γράψετε. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα διότι κάναμε πάρα πολλή δουλειά για αυτό το θέμα και ε, θέλουμε να τα μοιραστούμε μαζί σας. Θα τα απαντήσω αντίστροφα. Ε, λανθασμένη χρήση. Σε πρόταση ασφάλισης είναι πολύ ε, περιορισμένη η δυνατότητα λανθασμένης χρήσης, διότι θα είναι 18 ή 28 διαφορετικά συστήματα, επομένω είναι λίγο δύσκολο να υπάρξει τέτοιο πρόβλημα. Η δημιουργία του Ταμείου θεωρούμε ότι θα πρέπει να συμβαδίζει με κάποιο συντονισμό ή εναρμόνιση, να υπάρχουν κατάλληλα μέσα ελάχιστη έστω εναρμόνισης, διότι έχουμε διαπιστώσει ότι τα εθνικά ε, συστήματα επιδομάτων ε, ανεργίας ε, δεν μπορούν να να συντανιστούν, διότι σε κάποιες περιπτώσεις είναι υψηλότερα και σε κάποιες άλλες λιγότερα. Όσον αφορά τα υπάρχοντα κονδύλια, σίγουρα δεν επαρκούν. Ε, ταμεία όπως το Κοινωνικό Ταμείο ή το Ταμείο ε, Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, στόχο έχουν να αντιμετωπίσουν διαρθρωτικά ζητήματα, αναδιάρθρωση μεγάλων επιχειρήσεων, για παράδειγμα, σε περίπτωση μεταγκατάστασης. Ε, αυτό που προτείνουμε εμείς εδώ είναι αντίθετα να αντιμετωπίσουμε κυκλικά προβλήματα. Επομένως ε, δεν ε, υποκαθιστούνται, είναι συμπληρωματικά των ε, προβλημάτων αυτών. Και κάτι τελευταίο για το κόστος της μη Ευρώπης. Εμείς θεωρούμε ότι το κόστος της μη Ευρώπης είναι πολύ ψηλό ιδιαίτερα σε καταστροφικά γεγονότα, όπως για παράδειγμα η μεγάλη ύφεση, τα τελευταία δέκα χρόνια ή η ύφεση που είχαμε στις αρχές της δεκαετίας του 90 που έπληξε όχι μόνο τον Νότο αλλά και την ε, Βόρεια Ευρώπη και εμείς θεωρούμε ότι η επανασφάλιση μεταξύ των εθνικών ε, ταμείων είναι η κατάλληλη οδή, διότι δεν θα καλύψει τα συνηθισμένα, διότι λίγο πολύ τα κράτη-μέλη έχουν κράτος πρόνοιας που μπορεί να καλύψει τις βασικές ε, κρίσεις, αλλά θέλουμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ μεγάλη ύφεση όταν ταυτόχρονα υπάρχει και ανεργία και οι εθνικές αγορές ε, και ε, ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός έχουν περιορισμούς, επομένως ε, η πρόκληση να περιοριστούν τα επιδόματα ενεργείας όταν τα χρειαζόμαστε περισσότερο είναι πάρα πολύ μεγάλη και αυτό δεν θα πρέπει να γίνει και γι' αυτό ε, δεν θα πρέπει να έχουμε περιφερειακό πρόγραμμα, αλλά ευρωπαϊκό. Ευχαριστώ. Ε, λυπάμαι που δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερο χρόνο και δεν μπορώ να δώσω και περισσότερο χρόνο σε όλους όσους θέλουν να θέσουν ερωτήσεις, διότι Έχουμε ένα ακόμα σημείο στην ημερήσια διάταξη που πρέπει οπωσδήποτε να συζητήσουμε σήμερα. Επομένως σας ευχαριστώ όλους και για την ε, δέσμευσή σας και για τα αποτελέσματα που μας παρουσιάσατε. Κυρία Μασέλη, κύριε Ντάν, κύριε Νόιμεν και κύριε Μόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Ε, το κείμενο και τα στοιχεία τα έχετε στη διάθεσή σας, τα είδατε νωρίτερα. Μπορείτε να τα βρείτε όλα στην εφαρμογή e-meeting. Μπορείτε λοιπόν κάλλιστα να δείτε τα στοιχεία εάν θέλετε να εμπαθύνετε στα θέματα αυτά. Αλλά δεν μπορούμε να αφιερώσουμε εμείς περισσότερο χρόνο στο θέμα αυτό. Θα προσπαθήσουμε να επανέλθουμε με κάποιον άλλο τρόπο ίσως. Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν που ήρθατε εδώ σήμερα και που ε, κάνετε όλη αυτή τη δουλειά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ε, τώρα να πάμε στο σημείο 11 της ημερήσιας διάταξης. Η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την ενίσχυση της συνεργασίας ε, για την πρόληψη και αποτροπή της αδήλωτης εργασίας. επειδή υπάρχουν πιέσει από πλευράς χρόνου, θα ήθελα να ζητήσω σε όλους όσοι έχουν έρθει για το θέμα αυτό, να κάνετε σύντομες εισαγωγές. Καλώς ορίσατε. Θα έχετε τέσσερα λεπτά ο καθένας για την εισαγωγή σας. Και θα ξεκινήσω αν έχω σωστά τις πληροφορίες, με την κυρία Μιούρελ Γκίν από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εφόσον δεν έχω παρά μόνο τέσσερα λεπτά, να θυμίσω ότι προτείναμε και παρουσιάσαμε την πρόταση αυτή ήδη τον Ιούλιο, οπότε δεν θα επανέλθω επί των, με λεπτομέρειες επί της πρότασης αυτής. Αυτό που ήθελα να υπογραμμίσω τώρα είναι τρία σημεία. Καταρχήν, πιστεύω πως υπάρχει τώρα μία σύγκληση όσον αφορά τη συμφωνία, ε, όσον αφορά μάλλον ε, πολύ σημαντικές επιπτώσεις ανάμεσα στις οικονομικές και κοινωνικές ε, επιπτώσεις της μη δηλωμένη εργασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα όσον αφορά τη σημερινή διαχείριση και έξοδα από την κρίση αντίκτυπος για τι συνθήκε εργασία, υγεία και ασφάλεια, τα εργασιακά δικαιώματα όπως τα αναφέραμε προηγούμενα για τα επιδόματα κτλ. Αλλά και όσον αφορά τις προοπτικές συνταξιδότηση, την θεμητή, θεμητό ανταγωνισμό ανάμεσα στις εταιρείε και βεβαίω και το θέμα της μείωση των ε, φορολογικών εσόδων. Ε, επίσης, κοινωνικά ζητήματα όπως ας πούμε απασχόληση των γυναικών που επηρεάζονται πολύ από το φαινόμενο της μη δηλωμένης εργασίας και να θυμίσω ότι ε, όταν έγινε το τελευταίο η τελευταία δημοσκόπηση του Ευρωβαρόμετρου, Ένα στους δέκα, δήλωσαν ότι έχουν αγοράσει αγαθά ή υπηρεσίες που προέρχονται από μη δηλωμένη εργασία και ότι 4% των ανθρώπων επίσης είπαν ότι είχαν δουλέψει αδήλωτοι την προηγούμενη χρονιά. Δεύτερη παρατήρηση είναι να θυμίσω τους λόγους που οδήγησαν στην υποβολή αυτής της πρότασης. Ανάγκη για μια νέα μορφή ευρωπαϊκής συνεργασίας. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα τα οποία έχουν εφαρμοστεί εδώ και πολλά χρόνια ανάμεσα στα διάφορα μέλη και από διάφορου εμπειρογνώμονε. Η Κομισιόν έχει επίση χρηματοδοτήσει πολύ ενδιαφέροντα προγράμματα. Δεν ξεκινάμε από το μηδέν, ωστόσο έχουμε διαπιστώσει πω ε, υπήρχαν αρκετέ ελλείψει σε σχέση με τι δράσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως ε, τελείωσαν ανεπαρκή συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη γιατί διότι διαπιστώνουμε απουσία συνολικής σφαιρικής προσέγγισης, δηλαδή αν υπάρχουν κάποια κρατημέλη τα οποία εργάζονται με κάποιες καλές πρακτικές σε αυτό το τομέα, βλέπουμε ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης οι επιθεωρητές εργασίας, αυτοί που ελέγχουν δηλαδή την κοινωνική ασφάλιση, τα τελωνία, οι αρχές που ασχολούνται με τη μετανάστευση. Οι φορολογικέ αρχέ σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν συνεργάζονται μεταξύ του. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια πλατφόρμα που να τους επιτρέπει να συνεργαστούν. Δεν συγκεντρώνουν τι εμπειρίε τους και δεν τι ανταλλάσσουν. Και ένα άλλο τομέα, ένα άλλος παράγοντας μάλλον, είναι η δυσκολία των εθνικών αρχών και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να καλύψουν τις ε, διασυνοριακές ε, ε, πτυχές της μη δηλωμένης εργασίας. Παραδοσιακοί μηχανισμοί υπάρχουν για τις εθνικές πτυχές της μη δηλωμένης εργασίας. δεν υπάρχει αρκετή γνώση του πλαισίου άλλων κρατών μελών και υπάρχουν δυσκολίες ανταλλαγής πληροφοριών. Η πλατφόρμα λοιπόν που προτείνει η Κομισιόν σκοπεύει να καλύψει αυτές τις δυσκολίες και τα ελλείμματα. Τρίτο στοιχείο που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι είναι σαφές ότι στο πλαίσιο αυτής της νέας μορφής συνεργασίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να δουλέψουμε με διάφορους φορείς. Στο επίπεδο των εθνικών αρχών, όπως σας είπα και προηγουμένως, να εργαστούμε με διάφορα σώματα ελέγχου και πρόληψης και σε διάφορους τομείς, αλλά είναι εξίσου σημαντικό να ε, συνεργαστούμε με κοινωνικούς εταίρους που σε ορισμένα κράτη-μέλη συνεργάζονται άμεσα με τις ε, ελεγκτικές αρχές και τις αρχές πρόληψης. Υπάρχουν διάφορες καλές πρακτικές που εντοπίζονται στα διάφορα κράτη-μέλη και πρέπει να ε, συνεργαστούμε βεβαίως και με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν αναπτύξει εμπειρογνωμοσύνη εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και που μπορούν να επιτρέψουν στις δραστηριότητε της πλατφόρμας να ξεκινήσει τις εργασίες στις καλές προϋποθέσεις. Το... Ο οργανισμός της Λισαβόνας για την υγεία, ο, το Διεθνής Οργανισμός Εργασίας, με τον οποίο έχουμε ξεκινήσει κάποια συνεργασία ή με τις συνεργασία με τις επιθεωρήσεις εργασίας στα διάφορα κράτη-μέλη και αυτό είναι ένα κλειδί για την καλή συνεργασία να δουλέψουμε με πιο ολοκληρωμένο τρόπο. Αυτό αντικατοπτρίζεται στις προτάσεις μας από το γεγονό, με το γεγονός ότι ζητάμε από τα κράτη-μέλη να έχουν interface πολύ πιο συντονισμένο και γι' αυτό είναι και σημαντικό το να έχουμε συγκεκριμένα σημεία επαφής. Τελειώσαν τα τέσσερα λεπτά μου να υπογραμμίσω ότι το κλειδί για την καλύτερη στρατηγική θα ήταν ένα συνδυασμός μιας ενισχυμένης συνεργασίας σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Thank Σας ευχαριστώ πολύ και θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Μενάντες Βάλτε, που είναι ο διευθυντής ε, του Eurofund. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ που μας δίνετε στο Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη βελτίωση των συνθήκων ζωής και εργασίας σε το λόγο. Εργαστήκαμε σε αυτό το τομέα της αδήλωτης εργασίας, όπως και στο τομέα της εμπορίας και άλλους τομείς. Και οι δύο εκθέσεις που ε, μας προσέφεραν περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την πολιτική συζήτηση οδήγησαν στην βάση δεδομένων για τα μέτρα καταπολέμησης της μη δεδηλωμένης εργασίας. Έχουμε 186 μέτρα που προτείνουμε για καταπολέμηση της παράνομης εργασίας, της αδήλωτης εργασίας σε 33 χώρες, ανταλλαγή καλών πρακτικών που προσπαθεί να δείξει τι έχει ήδη δοκιμαστεί ε, στα κράτη-μέλη και βεβαίως οι αξιολογήσεις αυτές υπάρχουν για να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα. Αυτό το εργαλείο υπάρχει online και μπορεί κανείς να το εξετάσει ένα χώρο, ένα τομέα, ένα ομάδα στόχο, αλλά και ένα είδος μέτρου. Εξετάζουμε λοιπόν τα διάφορα είδη μέτρων εδώ, όχι μόνο τα παραδοσιακά, αλλά δηλαδή επιθεωρήσεις, ε, εντοπισμός και ποινές, αλλά και τα διορθωτικά μέτρα ε, για να μπορέσουμε να αυξήσουμε τη δέσμευση. Δηλαδή προσπαθούμε να δελάξουμε την παραδοσιακή στρατηγική του ε, της απειλής με την ε, πρακτική του κινήτρου για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε το επίπεδο. Είδαμε κάποια αλλαγή στις πρακτικές που χρησιμοποιούνται από τα κράτη-μέλη τα τελευταία χρόνια και από τις υποψήφιες χώρες ε, που έχουμε μελετήσει. Τα βασικά μέτρα είναι οι ποινές αλλά έχει υιοθετηθεί και μια μεγαλύτερη ε, ποικιλία μέτρων για να μπορέσουμε να ε, δούμε ποια, ε, ποια, ποια είναι η επιρροή των μέτρων αυτών. Τα βασικά διδάγματα που αποκομίσαμε είναι καταρχήν ότι το πρόβλημα είναι διαφορετικό σε μέγεθος ανάλογα με το κράτος μέλος πιο σημαντικό είναι ότι το προφίλ του μη διαδηλωμένου εργαζόμενου είναι διαφορετικό. Για κάποιες χώρες ε, οι μη δεδηλωμένοι είναι οι άνεργοι εργαζόμενοι, αλλά για κάποιες άλλες όχι. Είδαμε ότι δεν, υπάρχει μεγάλη δεν δίνεται μεγάλη προσοχή στη δέσμευση, αλλά περισσότερο στη συμμόρφωση. Και έχουμε συγκρίνει αυτά που υπόθηκαν, ότι δηλαδή τι γίνεται στα διάφορα επίπεδα. Δηλαδή δεν υπάρχει μεγάλη ανταλλαγή ε, ε, καλών πρακτικών. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρξει ανταλλαγή μέτρων πολιτικής όπου θα αξιολογηθεί ο στόχος κάθε μέτρου για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε κοινέ μονάδες για την αξιολόγηση. Και είναι σημαντικό να καταλάβουμε ποια μέτρα πολιτικής και ποιο συνδυασμός αυτών η ποια συχνότητα αυτών είναι η πιο αποτελεσματική στις διάφορες χώρες. Έχοντας τα όλα αυτά υπόψη, πιστεύουμε πως η πρόταση της Κομισιόν είναι καλή γιατί εστιάζει στην πρόληψη και την ε, αποτροπή της μη διδηλωμένης εργασίας, ιδιαίτερα όσον αφορά την ε, βελτίωση της, ε, της ενημέρωσης για τα διάφορα εργαλεία. Έχουμε ένα πρόγραμμα για το 2015 όπου θέλουμε να μπορέσουμε να μετατρέψουμε την βάση δεδομένων σε βάση δεδομένων που θα μπορεί κανείς να ενημερωθεί για να μπορούμε έτσι να έχουμε πιο εύκολη ανταλλαγή ε, των καλύτερων πρακτικών. Ζητούμε καλύτερο συντονισμό χωρίς παράταση της εντολής, δηλαδή έτσι λέμε ότι δεν έχουμε λεφτά ούτε για αυτό εδώ πέρα. Αυτό που αναμένεται είναι να παρακολουθεί κανείς τις συνεδριάσεις και να στέλνει τις διαθέσιμες πληροφορίες. Υπάρχουν επίσης κάποιες απόψεις ε, για να ολοκληρώσουμε στη διάρκεια της διαβούλευσης σε αυτό το κοινοβούλιο. Κάποιες, κάποιοι πρότειναν ότι η πλατφόρμα θα πρέπει να εντάσσεται στη Eurofarm. Πιστεύω που κάποιες φορές αυτό είναι σωστό, αλλά κάποιες φορές όχι. Και αυτό θα είναι καλύτερα να το δει η ίδια η Κομισιόν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και να δώσω το λόγο στον κύριο Τραμπ, ο οποίος εκπροσωπεί το, το Business Europe. Είσαστε λοιπόν ε, πρόεδρος της ε, Επιτροπής για τις ε, βιομηχανικές σχέσεις της, του Business Europe. Ευχαριστώ. Εκπροσωπώ το Business Europe, εκατομμύρια δηλαδή δηλωμένων επιχειρήσεων στην Ευρώπη που απασχολούν εκατομμύρια δηλωμένων εργαζομένων. Μας ανησυχεί λοιπόν το γεγονός ότι υπάρχει αθέμητος συνταγωνισμός επειδή υπάρχουν τόσοι αδήλωτοι εργαζόμενοι και τόσες αντίλατες επιχειρήσεις. Καλωσορίζουμε λοιπόν την πρόταση να δημιουργηθεί μια τέτοια πλατφόρμα. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να πιστεύουμε ότι αυτό θα αποτελέσει μια αυτόματη λύση. Να περάσω σε πιο συγκεκριμένους στόχους, οι οποίοι θεωρώ ότι λείπουν από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καταρχάς, και να αναφέρω αυτά που είπε το 2014 σε ψήφισμά του τον Γενάρη το Κοινοβούλιο, ότι δεν αρκεί να εφαρμόζονται κυρώσεις και να υπάρχει πιο πολλή συνεργασία μεταξύ των αρχών. Αυτό ασφαλώς είναι κάτι το καλοδεχούμενο, αλλά θα πρέπει να δημιουργηθεί και ένα γενικότερο περιβάλλον όπου δεν είναι τόσο κοστοβόρο το να είναι κανεί δηλωμένο είτε ω εργαζόμενος είτε ω εργοδότης στην Ευρώπη και να μην είναι τόσο εύκολο να είναι κανείς αντίλατος. Όσο λοιπόν δεν υπάρχει αυτή η ισορροπία πάντα θα είναι υπερβολικά μεγάλος ο αριθμό των αντίλατων στην Ευρώπη. Κατά δεύτερον, και αυτό θεωρώ ότι λείπει από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπή. Ναι, η πλατφόρμα θα πρέπει να αναλύει την κατάσταση στην Ευρώπη, αλλά δεν διευκρινίζεται τι είδου ανάλυση χρειάζεται θα θέλαμε λοιπόν να αναλύετε το γιατί σε κάποια κρατημέλη, σε κάποιες περιοχές είναι καλύτερο το περιβάλλον και οι πιο πολλές επιχειρήσεις είναι δηλωμένες και είναι μειονότητα αυτές που είναι αδήλωτες. Είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να διδαχτούμε από τα φωτεινά αυτά παραδείγματα και αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να το περιλαμβάνει η εντολή της πλατφόρμας, την ανάλυση των στοιχείων αυτών. Κατά δεύτερο, όπως αναφέρθηκε, προτείνεται να δημιουργηθεί μια βάση γνώσεων, βάση διμερών εμ, συμφωνιών. Προφανώς θα πρέπει να γίνονται τέτοιες διμερείς συμφωνίες, οι οποίες και θα πρέπει να δημοσιεύονται. Είναι λοιπόν πάρα πολύ δύσκολο να εξευρεθεί αυτή η ισορροπία στις συμφωνίες αυτές. Είναι καταπήγον το θέμα αυτό. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε την πλατφόρμα να καταστεί λειτουργική. Θα πρέπει να καλέσουμε τα κράτη-μέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να καταχωριστούν όλες αυτές οι δεμερείς συμφωνίες. Όλοι μπορούμε να εμπνευστούμε και να μάθουμε από αυτές. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε δύο χρόνια. Τέλος, ε, σε ό,τι αφορά την ψευδοαπασχόληση. Συμφωνούμε ότι αυτού του είδους η αυταπασχόληση θα πρέπει να καταπολεμηθεί ιδιαίτερως. Είναι μια απειλή μεγάλη για τις σωστές επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι αν το βάλουμε στην πλατφόρμα αυτή θα καθυστερήσει τη δράση, γιατί η ψευδοαπασχόληση είναι δηλωμένη απασχόληση. Τη γνωρίζει η αρχή του κάθε κράτους δεν θα πρέπει να μας καθυστερήσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπογραμμιστεί αυτό και τέλος ναι, να συμπεριληφθεί λοιπόν στην πλατφόρμα αλλά να μην αποτελέσει αυτό δικαιολογία για καθυστήρηση της πλατφόρμας γιατί οι αρχές γνωρίζουν ότι υπάρχει αυτή η απασχόληση, αυτή η ψευδής αυτοαπασχόληση. Αυτές λοιπόν ήταν οι συγκεκριμένες προτάσεις που είχα να κάνω. Ευχαριστώ. Ε, thank you. I'll... Ευχαριστώ. Η κυρία Γουόρνεκ, νομική σύμβουλος του Συνδικάτου ETUC. Σας ευχαριστώ πολύ. Το ETUC καλωσορίζει αυτή τη νέα ανεξάρτητη πλατφόρμα για την αδήλωτη εργασία και θέλουμε να γίνει υποχρεωτικό για όλα τα κράτη-μέλη και να υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση. Δεν είναι δυνατόν να σταματήσουμε ε, τη συνεργασία αυτή στην ανταλλαγή πληροφοριών και τις βέλτιτες πρακτικές. Θέλουμε καλύτερη εφαρμογή των υφιστάμε, του εφιστάμενου εργασιακού δικαίου. Χρειαζόμαστε καλύτερο συντονισμό, συγκεκριμένα μέσα, μέσα και υπάρχουν παραδείγματα και στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις επιθεωρήσεις εργασίας. Αν δείτε για παράδειγμα την έκκληση για την εισαγωγή μιας οδηγίας για κάποια ελάχιστα πρότυπα για τις επιθεωρήσεις και επίσης πρέπει να εφαρμοστούν συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής για την εκπαίδευση του προσωπικού και την κατάρτιση και να υπάρχουν κοινέ δράσεις ελέγχων για να καταπολεμήσουμε και τη διασυνοριακή αδήλωτη εργασία. Για το ETUC λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό όλα τα κράτη-μέλη να συμμετέχουν υποχρεωτικά σε αυτή τη νέα πλατφόρμα, αν όντω θέλουμε να έχουμε αποτελέσματα πανευρωπαϊκά. Και βεβαίως δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη νομική βάση ως ε, αιτιολογία για ε, χαμηλές προσδοκίες. Οι εκπρόσωποι των κρατών μελών στην πλατφόρμα θα πρέπει να έχουν και εντολή για το έργο τους στη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Αυτό προκειμένου η εργασία να είναι πραγματικά αποτελεσματική. Και βεβαίως για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και οι κοινωνικοί εταίροι σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε εθνικό επίπεδο να συμμετέχουν. Και αυτό ε, λόγω και του συγκεκριμένου ρόλου που έχουν να διαδραματίσουν. Όπως αναφέρθηκε ε, σε εθνικά συστήματα η ε, φορείς αυτοί έχουν διαδραματίσουν, οι κοινωνικοί εταίροι έχουν να διαδραματίσουν συγκεκριμένο ρόλο ε, και ο κοινωνικός διάλογος είναι αυτός ο οποίος θα βοηθήσει στην ε, πάταξη της αδήλωτης εργασίας. Ε, θα πρέπει να προστατεύονται επίσης και όσοι εργάζονται χωρίς να είναι δηλωμένοι, διότι αυτοί είναι τα πρώτα θύματα και μπορεί να, να δημιουργηθούν προβλήματα και παράνομες καταστάσεις. Προκειμένου λοιπόν να αλλάξουν τα πράγματα, θα θέλαμε να συσταθεί αυτή η πλατφόρμα με έμπνευση ε, της Επιτροπής ΣΛΙΚ, ε, διότι εκεί πραγματικά υπήρχε ε, εμπειρία από τη συνεργασία. Όσον αφορά τη συνεργασία θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η πλατφόρμα μπορεί να εργαστεί ανεξάρτητα και επομένως προτείνουμε να υπάρχει πρόεδρος και αντιπρόεδρος που θα εκλέγονται μεταξύ των μελών της πλατφόρμας και θα υπάρχει ένα ετήσιο πρόγραμμα και κατάλληλες εκθέσεις. Θα θέλαμε επίσης η Slick να είναι παρατηρητή στην πλατφόρμα, ώστε να συνδεθούν όλες οι υφιστάμενες δομές και προσπάθειες. Και προτείνουμε οι κοινωνικοί εταίροι να γίνουν μέλη, ώστε να μπορέσουν να διαδραματίσουν και αυτοί το ρόλο τους, όπως σας είπα προηγουμένως θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει σαφέστατη διάκριση μεταξύ εθνικής αδήλωτης εργασίας και διαμεθοριακής αδήλωτης εργασίας και ότι θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα καθήκοντα που θα σχετίζονται με τα δύο αυτά, ώστε να υπάρχει κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη και να υπάρχουν και κοινέ επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της διασυνοριακής ε, αδήλωτης εργασίας. Θα πρέπει να υπάρχει ένα αξιόπιστο και ταχύτατο σύστημα ανταλλαγή πληροφοριών, γιατί πολύ συχνά οι εθνικέ αρχέ χρειάζονται πολύ γρήγορα πληροφορίε από κάποιο άλλο κράτο μέλο. Το σύστημα IMI που αναφέρεται στο κείμενο είναι θεωρητικό σύστημα, που μάλιστα για μας υπάρχουν ερωτηματικά. Όσον αφορά το σημείο επαφής, θεωρούμε ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλες οι αρμόδιες αρχές συμμετέχουν ενεργά και ε, να υπάρχει και συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και επομένω θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία και να ε, συνοδεύουν όλοι το έργο αυτό. Μια τελευταία μου παρατήρηση, είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να καλύπτονται και οι αυτοαπασχολούμενοι. Αλλά στο κείμενο δεν αναφέρεται αυτό ούτε στου τόσκου ούτε στα καθήκοντά μα και αυτό θα πρέπει να προσθεθεί. Γι' αυτό ακριβώς και εμείς θέλουμε να έχουμε ένα πολύ ισχυρό κείμενο και να υπάρχει και πολύ φιλοδοξία στην εφαρμογή στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Τελευταίος ομιλητής, ο κύριος Τουσάν, πρόεδρος του ΣΛΙΚ, το οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως, που σημαίνει η Επιτροπή ε, Επιθεωρητών Εργασίας. Ε, ε ασχολείται μεταξύ άλλων και με την αδήλωτη εργασία. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την πρόσκληση αισθάνομαι μεγάλη τιμή. Ε, πρόκειται για... Ε, είμαστε το Ευρωπαϊκό Όργανο Επιθεώρησης Εργασίας ε, και εκπροσωπούνται όλοι οι εθνικοί οργανισμοί και συνεδριάζουμε δύο φορές το χρόνο με συγκεκριμένες θεματικές ασχολούμαστε. Έχουμε μια ολομέλεια όπου όλα τα κράτη-μέλη αντιπροσωπεύονται από κάποιον ε, εκπρόσωπο. Υπάρχουν διάφορες ομάδες εργασίας. Εγώ προσωπικά είμαι ε, πρόεδρος της ομάδας εργασίας παρατηρητήριο που αποτελεί τη σύνδεση ανάμεσα στο τομέα του εργατικού δικαίου και της ασφάλειας και ε, μας ζητήθηκε να ασχοληθούμε με τη δημιουργία αυτής της νέας πλατφόρμας για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. Καταρχήν στη σύστασή μας, την οποία διατυπώσαμε, ήμασταν της άποψης ότι θα πρέπει καταρχήν να εκμεταλλευτούμε, γιατί υπάρχουν διάφορες πλατφόρμες που ήδη υπάρχουν όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών που έχουν δημιουργηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο Κάποιες φορές μάλιστα με περιορισμένη συμμετοχή ορισμένων κρατών, όπως ας πούμε Σύμπλες ή το ISLNU ή άλλες πλατφόρμες. Πρέπει δηλαδή να εκμεταλλευτούμε στο maximum τις υπάρχουσες βάσεις, αντί να δημιουργήσουμε ακόμα μία πλατφόρμα. Θα πρέπει να δώσουμε δηλαδή ένα καλό παράδειγμα εργασίας του SLIC της Επιτροπής που είναι υπεύθυνη ε, για τις επιθεωρήσεις εργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να δώσει ένα καλό παράδειγμα με όλες τις ομάδες εργασίας που έχει δημιουργήσει και ίσως ε, το μόνο μειονέκτημα είναι ότι θα είναι πιο περίπλοκο γιατί εδώ έχουμε τις υπηρεσίες επιθεώρησης εργασίας που είναι μέλη ε, ούτως ή άλλως δηλαδή κανονικά υπηρεσίες επιθεώρησης εργασίας που είναι υπεύθυνες στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας εδώ θα είναι πιο περίπλοκο γιατί είναι πιο πολλοί οι παράγοντες τουλάχιστον στο επίπεδο των θεσμών, στο κράτη-μέλη δηλαδή, όπου έχουμε φυσικά τις υπηρεσίες επιθεώρησης, εργασίας, επίσης τις υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης αλλά και τις υπηρεσίες φορολόγησης και μιλώ τις εφορίες και μιλώ για ε, τις κρατικές ε, τις, ε, τους κρατικούς θεσμούς. Πρέπει να δούμε επίσης ε, και για δημοσιονομικούς λόγους πώς θα συνεδριαστούμε. Δύο μέλη καλούνταν. Τώρα με την επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, περιοριζόμαστε σε έναν εκπρόσωπο αναχώρα. Υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα με την συμφωνία της Προεδρίας να σταλεί κάποιος παρατηρητής ή ένας εμπειρογνώμονας ένα θέμα. Γιατί Μπορεί να χρειαστεί, να μην έχει κανείς δηλαδή απόλυτη γνώση όλων των τομέων που συζητώνται κάθε φορά. Πάντως, σε κάθε συνεδρίαση έχουμε ατζέντα εξαιρετικά καλά οργανωμένη εκ των προτέρων με κατάσταση πρόοδου για κάθε ομάδα εργασίας για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε τα θέματα που υποβάλλονται στο ΣΛΙΚ. Έχουμε ομάδες εργασίας για τον έλεγχο, για την ε, επιβολή των νόμων. Έχουμε ομάδες εργασίας όπου εκπροσωπούνται όλες οι ομάδες εργασίας και σε άλλες περιπτώσεις γίνεται επί τη βάση ομάδα εργασίας όσον αφορά τις εργαλειομηχανές, τις επικίνδυνες ουσίες, την διασυνοριακή επιβολή και η τελευταία ομάδα εργασίας που δημιουργήθηκε ήταν το παρατηρητήριο. Οι εκθέσεις μας ε, δημοσιεύονται για το, στο σύνολο των μελών ε, που μπορούν να σχολιάσουν και όσον αφορά τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν πάντοτε λαμβάνονται στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ που με επιτρέψατε να πάρω το λόγο. Thank you for your <clears throat> introduction. Σας ευχαριστώ για τις εγωγές αυτές. Και τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Πρίνσκι από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες που είναι υπεύθυνος για την έκθεση την οποία επεξεργαζόμαστε εδώ στα πλαίσια του Κοινοβουλίου. Thank you, Madam Chair. Permit me first of all to express... Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να εκφράσω την εκτίμησή μου για τις παρουσιάσεις που μόλις ακούσαμε. Όλοι κατανοούμε πόσο περίπλοκο είναι το πρόβλημα της ε, αδήλωτης εργασίας και του ότι χρειάζεται μια πραγματικά συντονισμένη απάντηση από διάφορες πλευρές. Η πλατφόρμα η οποία προτείνεται λοιπόν από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταδεικνύει το πρόβλημα που αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί πάντως ε, μία πρόκληση προκειμένου τον εργαλείο αυτό να καταστεί ένα μέσο προστιθέμενης αξίας και όχι ένα μέσο το οποίο θα επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν, Πρόεδρε, θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα. Και αν θα μπορούσαν ε, όλοι όσοι πήραν το λόγο να σχολιάσουν και μετά θα προσπαθήσω να επικεντρώσω το ερώτημα πιο συγκεκριμένα. Το γενικό ερώτημα. Θα ήταν ωφέλιμο και χρήσιμο να προσπαθήσουμε να ορίσουμε με συγκεκριμένο τρόπο την ακριβή φύση του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε και εξηγούμε. Στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται και είναι το πρώτο κείμενο αυτό στο, στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τι είναι η αδήλωτη εργασία. Οποιαδήποτε ε, δραστηριότητα ε, επιπληρωμή νόμιμη ως προς τη φύση της, αλλά όχι δηλωμένη στις δημόσιες αρχές. Το ερώτημα λοιπόν που ανακύπτει είναι το εξής. Το πρόβλημα της αδήλωτης εργασίας, μάλλον η αδήλωτη εργασία, είναι πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν καταγράφεται, το οποίο δεν το καταγράφουν οι δημόσιες αρχές. Το θέτω λοιπόν το ερώτημα αυτό, γιατί το θέμα της αδήλωτης εργασίας έχει να κάνει με τη ζήτηση νόμιμων δραστηριοτήτων και με την, με την ε, ύπαρξη προσφοράς. Είναι λοιπόν δραστηριότητε τι οποίε οι επιχειρήσει ενδιαφέρονται να έχουν και τι οποίε ενδιαφέρονται να δώσουν οι εργαζόμενοι. Το γεγονό ότι είναι αδήλωτη αυτή η εργασία δε, έχει πολύ σοβαρέ επιπτώσει και για του εργαζόμενου που εργάζονται υπό επισφαλεί όρους και έχουν πολύ λιγότερη προνόμια και σε ό,τι αφορά τον αθέμητο ανταγωνισμό, σε ό,τι αφορά τις τοπικές κοινωνίες, σε ό,τι αφορά τις δημόσιες αρχές, όλες τις εισφορές που χάνονται. Θεωρώ λοιπόν ότι οι προκλήσεις ε, που θα αντιμετωπίζουμε στην πλατφόρμα αυτή θα είναι το πώς θα μπορούμε να βάλουμε στον νόμιμο κύκλο εργασιών την αδελαιότητα εργασία. Γιατί μιλάμε κατά πολέμηση της της εργασίας, πρόληψη, αποφυγή και το καθεξής. Ρωτώ λοιπόν καταρχάς το την κυρία Γκουέν. Σε ό,τι αφορά την ε, μη τηλεμένη εργασία. Συμφωνείτε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο μέλλον θα μπορούσε να εξετάσει πολύ σοβαρά τις δύο πτυχές, τις δύο, τα δύο πρόσωπα του προβλήματος. Καταρχάς, σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας για την αδέλετη εργασία, αλλά εκ παραλλήλου τα μέτρα τα οποία θα ενθαρρύνουν όσους απασχολούνται σε τέτοιο καθεστώς να δηλωθούν. Να τερθώσουν την κατάστασή τους. Και προς τον Αυτό το αξίωμα των κινήτρων και των ε, ποινών μπορείτε να μας το αναπτύξετε. Πώς μπορούμε δηλαδή να θέσουμε ε, εξίσου την έμφαση και στα θέματα εφαρμογής αλλά και στα θέματα ε, δυνατοτήτων που μπορούμε να δώσουμε στους εργαζομένους αυτούς. Προς την κύριε Τράμπε. Στον κύριο Τράμπε. Μας παρουσιάσατε επαρκώς ε, τις ανησυχίες των δηλωμένων επιχειρήσεων και όλες τις αρνητικές επιπτώσεις της αντίλωτης εργασίας. Ωστόσο, αναφερθήκατε και στην αρχή του ότι είναι πολύ ακριβή η δηλωμένη εργασία στην Ένωση. Θα θέλατε δηλαδή να μειωθεί η αδήλωτη εργασία και όχι να γίνει δηλωμένη εργασία, μιας και είναι τόσο υψηλός το κόστος. Πιστεύετε πραγματικά ότι αυτό είναι δικαιολογημένο, γιατί είτε είναι ακριβό είτε δεν είναι ακριβό το να είναι δηλωμένη εργασία, τουλάχιστον υπάρχει διαπραγμάτευση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, υπάρχει αξιολόγηση από πλευράς ε, των ε, ανταγωνιστών. Την κυρία Βάρνεκ τώρα. Από την ΕΤΟΚ. Από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εργαζομένων. Πείτε μας αν θέλετε, ποια είναι η εμπειρία σας έως τώρα για την νομιμοποίηση της αδήλωτης εργασίας από πλευρά συνδικάτων. Ποια είναι μια δικαιολογημένη στρατηγική που θα μπορούσε να ακολουθήσει η πλατφόρμα. και σε τι αφορά τους εργαζόμενους που είτε ηθελημένα είτε μη υπησέρχονται σε αυτό το κύκλο της αντίληπτης εργασίας. Ποιος θα ήταν λοιπόν ο ενεργός ο ρόλος σας μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους, με τις επιχειρήσεις, μαζί με τις αρχές, τι ευρωπαϊκές και τις εθνικές. Για αυτό το πολύ σοβαρό, περίπλοκο και επώδυνο πρόβλημα. Και τέλος να καλέσω τους συναδέλφους και όλους όσοι είναι στην αίθουσα να προσπαθήσουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να αποτελέσει αυτή η πλατφόρμα μια προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να είναι συλλογματική αυτή η προσπάθεια προς την προσπάθεια των κρατών μελών, των κοινωνικών εταίρων, τους ΛΙΚ και πολλών άλλων φορέων προκειμένου να υπάρξει και η αντίληψη ότι το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται σοβαρά και με συνέπεια. Ευχαριστώ. 25 λεπτά λέει η Πρόεδρος έχουμε ακόμα. Νομίζω ότι το πιο χρήσιμο θα ήταν να δώσετε λίγο πιο σύντομες απαντήσεις και οι πέντε του πάνελ και να δούμε στη συνέχεια αν υπάρχει χρόνος για παρεμβάσεις και από τα μέλη της Επιτροπής μας. Η κυρία Γκουίν, καταρχάς, αν μπορεί να ξεκινήσετε εσεί. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Για το θέμα αυτό της προσφοράς και της ζήτησης, ε, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αξιολόγηση επιπτώσεων που έκανε για να κάνει την πρόταση έλαβε υπόψη τη την πολύ σημαντική διάσταση του φαινομένου και το γεγονός ότι ε, προκύπτει σε διάφορα κράτη-μέλη για λόγους ε, πολυδιάστατους. Και θα πρέπει να τα δούμε και λίγο πιο προσεκτικά. Σαφέστατα η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δίνει προτεραιότητα σε μια μορφή συνεργασίας μεταξύ των αρχών των κρατών μελών επειδή δεν υπάρχουν ε, βήματα όπως ε, ανέφεραν και όσοι ε, αναφέρθηκαν στα θέματα αυτά και επειδή πρέπει να έχουμε πρόληψη και έλεγχο, δεν είναι μόνο έλεγχος αλλά είναι και η πρόληψη που μετράει, θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν ένα πιο συνολικό όραμα και μια καλύτερη ανάλυση του φαινομένου. Το θέμα της επισημοποίησης της εργασίας και της αδήλωτης εργασίας θα μπορούσε να εξεταστεί και από την ανταλλαγή ε, απόψεων για τα μέτρα που έχουν εφαρμόσει τα διάφορα κράτη-μέλη. Ε, αναφερθήκατε στο θέμα αυτό πριν από λίγο. Σαφώς, πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να ε, τονίσει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και φυσικά ε, των ε, απαραίτητων εταίρων για να έχουμε μια προστιθέμενη αξία σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως για παράδειγμα του κοινωνικού εταίρου, τις διάφορες υπηρεσίε κ.ο.κ. Αλλά βεβαίως κάποιες δραστηριότητες θα έχουν ε, σίγουρα ε, συνέπειες στην ανάλυση και στην ομιμοποίηση της αδήλωτης εργασίας και φυσικά και τις την ανάλυση των διαφόρων ε, βέλτιστων πρακτικών που υπάρχουν στα κάποια κράτη-μέλη. Ε, σε επίπεδο εθνικό επίσης θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο τα θέματα, να υπάρχει και κοινή εργασία και σε διεθνές επίπεδο, σε επίπεδο Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας ε, που κάνει μια σχετική μελέτη και θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματα του χρόνου για την άτυπη εργασία. Πρόκειται για κάτι το οποίο περιλαμβάνει κράτη που έχουν τελείως διαφορετικές εμπειρίες ε, ε, από τις εμπειρίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αλλά το φαινόμενο της νομιμοποίησης της αδήλωτης εργασίας είναι μεταξύ των θεμάτων της έκθεσης και θα υπάρχουν και κάποιοι κοινοί προσανατολισμοί σε διεθνές επίπεδο και στο σημείο αυτό. Ο κύριος Μενέντες Βάλτες αν κατάλαβα καλά, θέλετε κάποιες ε, περαιτέρω πληροφορίες για τις διαφορετικές ε, προσεγγίσεις, αυτές τις ε, ποινές και τα κίνητρα. όταν υπάρχει παράνομη δραστηριότητα θα πρέπει να υπάρχει κίνητρο, δηλαδή έχεις κάτι όφελο, ως ε, το οποίο υπερκερ, ε, ε, υπερτερεί αυτόν που έχεις να χάσεις και φυσικά θα πρέπει να υπάρχει και το ηθικό ζήτημα. Υπάρχουν διάφορες λοιπόν εκστρατείες οι οποίες αντιμετωπίζουν τα διάφορα στοιχεία του φαινομένου και έχουμε συλλέξει και διάφορα παραδείγματα επ' αυτού. Ωστόσο, και νομίζω ότι αυτό το επανέλαβε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, είναι πολύ σημαντικό να γίνεται αξιολόγηση. Αξιολογούνται πολλά, αλλά δεν έχουν αξιολογηθεί τα πάντα. Ε, δεν είναι συγκρίσιμες δυστυχώς οι αξιολογήσεις και μπορούμε να έχουμε ίσως ε, κάποιες κοινέ μονάδες αξιολόγησης, να βλέπουμε για παράδειγμα την αναλογία κόστους ωφελίας σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί για κάποιο συγκεκριμένο μέτρο ε, να προσπαθούμε λοιπόν να αντιληφθούμε ποια είναι τα πιο αποτελεσματικά μέτρα, αλλά επίσης και την κατάλληλη ακολουθία και το κατάλληλο πλαίσιο ώστε να είναι πιο αποτελεσματικά αυτά τα μέτρα. Ε, υπ' αυτή την έννοια η ανταλλαγή γνώσεων δεν είναι μόνο ανταλλαγή καλών πρακτικών, αλλά είναι ε, και ε, μια διαδικασία μάθησης που μας επιτρέπει να μάθουμε ποια είναι τα πιο αποτελεσματικά από πλευράς κόστους μέσα και αυτό είναι χρήσιμο, μπορεί να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα είναι πολύ δύσκολο να γίνει σε ατομικό επίπεδο από κάθε κράτος μέλος. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Ε, εμείς βεβαίως είμαστε ένα υπέρ της ενίσχυσης των ελέγχων. Αυτό θα μπορέσει να μας βοηθήσει να ε, μειώσουμε κάποια από τα προβλήματα της αδήλωτης εργασίας, αλλά θεωρούμε ότι αυτό πόρο απέχει από την επίτευξη του στόχου μας. Θα πρέπει να ε, δημιουργήσουμε κοινωνίες τις οποίες οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι όταν ε, εργάζονται νομίμως, πληρώνουν κοινωνική ασφάλιση και φορολογία, αλλά λαμβάνουν και κάτι ως αντάλλαγμα για όσα καταβάλουν βάση νομοθεσίας. Και βεβαίως υπάρχουν και τμήματα της Ευρώπης που έχουν καλύτερες επιδόσεις από άλλες περιοχές της Ευρώπης. Ε, χώρες στις οποίες θεωρείται φυσιολογικό να είναι κάποιος νομίμος ε, στη χώρα, εργάζεται, να εργάζεται νομίμος και να ε, καταβάλει τους φόρους τους και να πληρώνουν κοινωνική ασφάλιση. Αν θέλουμε λοιπόν να αναλύσουμε κάτι στην πρόταση, θα πρέπει να αναλύσουμε αυτό. Εάν μπορούμε να αντλήσουμε διδάγματα από άλλα κράτη-μέλη, ώστε να είναι πολύ χαμηλότερο το επίπεδο της αδήλωτης εργασίας, διότι μπορούμε να αντλήσουμε διδάγματα, θεωρώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Νομίζω ότι πριν ε, ε, πω την άποψή μου θα πρέπει να έχουμε ένα σαφή ορισμό του τι ακριβώς εννοούμε αδήλωτη εργασία, τη δηλωμένη εργασία και από εκεί και πέρα να δούμε τους δείχτες όσον αφορά τη δηλωμένη και την αδήλωτη εργασία. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο θα έπρεπε να μας απασχολεί είναι κυρίως ε, οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε επισφαλείς συνθήκες. Υπάρχουν εργαζόμενοι που είναι θύματα του ανταγωνισμού από άλλες, κάποιου οι οποίοι είναι αδήλωτοι και φυσικά υπάρχει και το κράτος το οποίο χάνει έσοδα διότι δεν ε, ε, καταβάλλονται εισφορές ε, για κοινωνική ασφάλιση, δεν καταβάλλονται φόροι. Εδώ σκέφτομαι ακόμα και τη βελγική κυβέρνηση, η οποία θα πρέπει να δει αν υπάρχουν και κάποιοι υπερβολικοί διοικητικοί φραγμοί όσον αφορά τον τρόπο δήλωσης της εργασίας. Αυτός είναι ο λόγος ίσως για παράδειγμα που στο Βέλγιο έχουμε επενδύσει το τελευταίο διάστημα ε, ε, στη διαβίβαση ε, με ηλεκτρονικό τρόπο των στοιχείων. Είναι μια μεγάλη διαδικασία όσον αφορά την καταγραφή των παρόντων στα εργοτάξια, διότι εμείς από πλευρά ΣΛΙΚ είμαστε βέβαιοι ότι η αδήλωτη εργασία δεν περιορίζεται μόνο στα σύνορα, αλλά ότι είναι ιδιαίτερα εφευρετικοί όσοι κάνουν αδήλωτη εργασία. Υπάρχουν, για παράδειγμα, Ε, δυνατότητα να ε, υπάρχουν εργοτάξια που χρησιμοποιούν ε, γραφεία προσωρινά απασχολούμενων και ο ένας σε στον άλλον και έτσι προχωράει η αδηλωτή εργασία. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Όσον αφορά τα συνδικάτα, ένα παράδειγμα είναι ότι τα συνδικάτα ούτως ή άλλως ε, προσπαθούν να ενημερώνουν καταλήλως τους εργαζομένους και πρώτη τους δράση είναι να τους ενημερώνουν για τα δικαιώματά τους και να τους λένε σε ποιες περιπτώσεις υπάρχουν καταχρήσεις και τι δικαιώματα έχουν σε κάθε κράτος μέλος. Υπάρχουν λοιπόν σωματεία τα οποία έχουν συσταθεί ακριβώς ε, για να δίνουν αυτές τις πληροφορίες στους εργαζομένους. Και όπως σας είπα και προηγουμένως, ο ρόλος των συλλογικών συμβάσεων ε, θα πρέπει να καλύπτει και τα θέματα της αδήλωτης εργασίας, διότι η έρευνα έχει καταδείξει, έρευνα για παράδειγμα του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, ότι τα επίπεδα των μισθών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά το επίπεδο αδήλα της εργασίας στα διάφορα κράτη-μέλη. Αν υπάρχουν καλές συλλογικέ συμβάσεις με αξιοπρεπέ επίπεδα μισθών και καλά επίπεδα μισθών, αυτό θα επηρεάσει και τον, το ποσοστό της αδήλωτης εργασίας. Γι' αυτό ακριβώς αναφέρθηκα στους ε, μηχανισμούς διαπραγμάτευσης των συλλογικών συμβάσεων ε, προηγουμένως. Ο ρόλος των συνδικάτων βεβαίως και αυτό φαίνεται και σε κάποια κράτη-μέλη περισσότερο, είναι να ελέγχουν τις συνθήκες εργασίας στις διάφορες επιχειρήσεις, ε, να έχουν τη θέση τους εκεί και για μας είναι πολύ σημαντικό για τα συνδικάτα να έχουν πρόσβαση στις επιχειρήσεις ακριβώς γι' αυτό το λόγο, για να μπορούν να δουν η διεισόμαση τι συμβαίνει επί τόπου. Και μια τελευταία παρατήρηση, διότι ρωτήσατε πώς μπορούμε να νομιμοποιήσουμε τους εργαζομένους που δουλεύουν αδήλωτοι. Εμείς θεωρούμε ότι θα ήταν ήδη πολύ χρήσιμο αν οι νομικοί συνέπειες σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχουν αδήλωτοι εργαζόμενοι εάν τους δίνονται όλα τα δικαιώματα ε, που ε, έχει ένας νόμιμα εργαζόμενος όταν νομιμοποιούνται, σίγουρα θα διευκολυνθεί η κατάσταση. Ε, η Πρόεδρος, υπάρχει κάποιος από τους σκιώδεις συζητητές εδώ στην αίθουσα που θα ήθελε να λάβει το λόγο από τους συντηρητικούς και δημοκράτες και από την Ευρώπη της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας και το ΕΛΚ εδώ. Μια σύντομη ερώτηση από το ΕΛΚ, μια σύντομη ερώτηση από την Ενωτική στερά, το FTD και από την κυρία Χάρκιν και από το ECR. Και η κυρία Κούνεβα φυσικά. Βεβαίω, Θα ξεκινήσουμε με την κυρία Κούνεβα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να, όμως δεν τα κάνω ερώτηση. Η η διασφάλιση, η των δικαιωμάτων των εργαζομένων είναι θέμα πολιτισμού μιας κοινωνίας. Δεν μπορεί να υπάρχει τεχνική και οικονομική πρόοδος εις βάρος της υγείας και της ασφάλισης των εργαζομένων. Οι πολίτες μας είχαν χρόνια να περάσουν τόσο δύσκολα όσον αφορά την διασφάλιση των κοινωνικών τους δικαιωμάτων και έχουν στραμμένα τα βλέμματα τους επάνω μας. Είναι πολύ σημαντικό ότι αποφασίσαμε να δούμε το πρόβλημα της αδέλφωσης εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό όμως πρέπει να είναι μόνο η αρχή Πράγματι, η ευρωπαϊκή συνεργασία και ανταλλαγή καλών πρακτικών θα βοηθήσει τις εθνικές αρχές τις δικές τους πολιτικές. Πρέπει όμως να υιοθετήσουμε όλοι συγκεκριμένους κανόνες πρόληψης και επιβολής για την μεγαλύτερη δυνατή προστασία και καταπολεμήσει το φαινομένο. Οι εργοδότες που διστάζουν να προχωρήσουν σε δεσμευτικά μέτρα αν δεν θέλουν να σκεφτούν την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων να σκεφτούν τον αθέμητο ανταγωνισμό που δημιουργούν κατά των σωστών επιχειρηματιών. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο τρόπο τη συμμετοχή των εργαζομένων στην πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί γιατί έχουμε να μάθουμε πολλά από την εμπειρία τους. Πρέπει να ορίσουμε πολύ προσεκτικά το καθεστώς του παρατηρητή που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρόταση της. Οι εργαζόμενοι πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά με προτάσεις. Το το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει λόγο στο πρόγραμμα που ορίζει η πλατφόρμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank uh, Εγώ σας ευχαριστώ και θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Ρουμάνα Τόμκ από το ΕΛΚ. Σύντομη ερώτηση μόνο. Αν ναι, είναι δυνατόν. Yes, Ένα σύντομο σχόλιο, αν μου επιτρέπετε. Σας ευχαριστώ για αυτή τη δυνατότητα που μου δίνετε να ε, μοιραστώ μαζί σας ε, κάποιες σκέψεις για αυτό το θέμα. Βεβαίως ε, χαιρετίζω όλους τους στόχους που έχουν τεθεί για τη μείωση της αδήλωτης εργασίας σε όλα τα κρατημέλη και καθώς και τις δυνατότητες που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην μείωση της ε, αδήλωτης εργασίας, δηλαδή την ανταλλαγή στοιχείων, αναλύσεων, καλών πρακτικών ανάμεσα στις χώρες μέλη. Ωστόσο, θεωρώ ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το εξής εάν θέλουμε να είμαστε επιτυχείς σε αυτή τη δραστηριότητα. Καταρχήν, πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας έναν ακριβή ορισμό της, εργασίας, της αδήλωτης εργασίας. Αν δεν έχουμε έναν τέτοιο ορισμό, ο στόχος θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Αλλά καταρχήν θα πρέπει επίσης να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν στην ε, εκδήλωση αυτού του φαινομένου, γιατί οι λόγοι αυτοί διαφέρουν από τη μια χώρα στην άλλη, αλλά είμαι πεπισμένος ότι, πεπισμένη ότι στις περισσότερες χώρες μέλη το βασικό αίτιο είναι η υπερβολική, το υπερβολικό φο, φόρτος που αραίνει την εργασία. Εάν θέλουμε λοιπόν να καταφέρουμε να απαλλαγούμε από την αδύνατη εργασία θα πρέπει να σκεφτούμε τρόπους ώστε να ε, προλάβουμε τα αίτια που οδηγούν σε αυτού του είδους την ε, απασχόληση. Τέλος, για να κλείσω, θα ήθελα επίσης να συμφωνήσω με τα όσα αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο, δηλαδή ότι οι εργαζόμενοι δεν θέλουν ε, πάντοτε να είναι ανεξάρτητοι, να δηλωθούν ως ανεξάρτητοι επαγγελματίε για να αποφύγουν ε, φορολόγηση. Πολύ συχνά οι ίδιοι εργοδότες είναι αυτοί που θέλουν να αποφύγουν μικτές αμοιβέ, μικτούς μισθούς εξαιρετικά υψηλούς και αναγκάζουν τους ε, εργαζόμενους τους να, να ανατρέξουν σε άλλες μορφές εργασίας, δηλαδή την εργασία ως ανεξάρτητοι επαγγελματίες. Αυτό το πρόβλημα λοιπόν θα πρέπει επίσης να εξεταστεί από διαφορετική άποψη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Χάρκιν, ECR. Μάκινταρ λέγομαι, αλλά εντάξει δεν πειράζει. Ε, θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τους εισηγητές που ακούσαμε σήμερα, καθώς επίσης τον εισηγητή μας. Ε, καλωσορίζω τις εξελίξεις Έσβησε το μικρόφωνο της ομιλήτριας. Καλωσορίζω λοιπόν αυτή την πρόταση για ανταλλαγή καλύτερων πρακτικών και πληροφοριών, καθώς και καλύτερη κατανόηση για την αδήλωτη εργασία. Υπάρχει ένας πολύ ξεκάθαρος ορισμός από την Κομισιόν ότι η αδήλωτη εργασία είναι οποιαδήποτε αμοιβόμενη δραστηριότητα που είναι νόμιμη στη φύση της αλλά δεν δηλώνεται στις δημόσιες αρχές. Ε, οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα είναι εκτός αυτού του πεδίου. Δεν μιλάμε για αυτές τις παράνομες, μιλάμε για τις νόμιμες δραστηριότητες που δεν δηλώνονται ωστόσο. είναι σοβαρό το θέμα γιατί έχει ε, αντίκτυπο σε όλα τα κρατη Είναι ένα πρόβλημα όσον αφορά την φοροαποφυγή και επίσης ε, την απάτη στα επιδόματα. Αλλά ε, Επίσης ε, προκαλεί αθέμητο ανταγωνισμό για τις επιχειρήσεις και τα άτομα που συμμορφώνονται προς την νομοθεσία και που ε, δηλώνουν σωστά τους εργαζόμενους τους. Η φύση και η κλίμακα της αδήλωτης εργασίας ε, δικημένεται από τη μια χώρα στην άλλη Οπότε μια ομοιόμορφη γενική προσέγγιση δεν θα λειτουργήσει. Ορισμένα θα ωφεληθούν πολύ περισσότερο από ό,τι άλλα από αυτήν την πλατφόρμα. Και θα πρέπει να πω ότι εγώ είμαι εδώ ε, αντιπροσωπεύοντας τα δυτικά Midlands ε, του Ηνωμένου Βασιλείου και θέλω να ε, εξασφαλίσω ότι θα πάρουμε τα λεφτά μας πίσω για τους φορολογούμενούς μας. Ξέρω ότι στη χώρα μου το μέγεθος αυτού του προβλήματος είναι πολύ μικρότερο από ό,τι σε άλλες χώρες. Οπότε ε, μου φάνηκαν ενδιαφέροντα αυτά που είπε η Business Europe να διευκολυνθεί η διαδικασία και να γίνει λιγότερο δαπανηρή για την δήλωση των εργαζομένων. Ξέρω ότι όταν έκανα μια σχετική εργασία έκθεση για αυτή την επιτροπή, σε κάποιε χώρε αυτό παίρνει τέσσερι μέρε, ενώ σε άλλε 40 για να δηλώσει κανεί έναν εργαζόμενο. Και αυτό σημαίνει μέγα κόστο. Ε, Βεβαίω η νομοθεσία, ο νόμος πρέπει να επιβληθεί, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ταυτόχρονα ότι είναι και σωστός και καλύτερη η νομοθεσία όπου γίνεται, ώστε ο κόσμος πιο εύκολα να μπορεί να συμμορφωθεί προς αυτήν. Γνωρίζω ότι υπάρχουν ε, ε, ανησυχίες που εκφράζονται κυρίως στο έγγραφο του Συμβουλίου για το ότι δεν έχουμε εξαντλητικό κατάλογο πρωτοβουλειών, ενώ ταυτόχρονα ε, αυτός είναι υποχρεωτικός. Δεν είναι λογικό να προτείνθει κάτι τέτοιο. Εγώ θα ήθελα να υπάρξει εθελοντική προσέγγιση ώστε να, μπορεί να μπορούν μάλλον όλοι να το υποστηρίξουν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ σχεδόν μας τελείωσε ο χρόνος. Η κυρία Τόν είναι εδώ από την Άλντε γιατί είναι η σκιώδης η Γιατί ήθελα να ακούσουμε πρώτα το σκιώδη. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να περάσουμε στη Μπεγκίν από το EFTD. Ευχαριστώ πολύ. Να μπω αμέσω στην ουσία αυτή τη πρόταση. κατά πολέμηση της ε, ε, δήλωτη εργασία είναι ένα δίκαιο και σημαντικό αγώνα για πολλέ χώρε και κυρίω για τη δική μου χώρα, που έχει μία από τι πρώτε θέσει ε, στην Ευρώπη όσον αφορά τον λόγο μεταξύ αδήλωτη εργασία και, και ΑΕΠ. Ακριβώς επειδή είναι τόσο σοβαρό το θέμα θα ήθελα να κατανοήσω αν τελικά είναι καλύτερη αυτή η επιλογή για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτόν τον αγώνα. Υπάρχουν πολλές διαφορές κράτη-μέλη και πολλά διεθνή φόρα ε, όπου συζητείται για δήλωτη εργασία, οπότε ο κίνδυνος επικάλυψης είναι εξαιρετικά υψηλός. Θα ήθελα να καταλάβω ποια είναι η προστιθέμενη αξία αυτής της πλατφόρμας, αυτής της βάσης, τι θα μπορούσε να μας προσφέρει, ποιο είναι το πλεονέκτημα για τους συμπολίτε μας, ε, ε, αν και είναι μικρό το κόστος για τον δημόσιο προπολογισμό θα πρέπει να ξέρουμε ποια είναι τα αποτελέσματα που επιθυμούμε και πόσο συχνά θα συνεδριάζουν οι συμμετέχοντες σε αυτή την ε, πλατφόρμα, ποιοι θα είναι, σε τι επίπεδο, εάν η Κομισιόν θέλει να προωθήσει την συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και ως μέλος και όχι ως παρατηρητή. Υπάρχουν πολλά ανοιχτά εκκρεμή θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν εις βάθος. Ελπίζω πως η Κομισιόν θα μπορέσει να απαντήσει στα ερωτήματα που έθεσα γιατί είναι σημαντικό να βρούμε συγκεκριμένη λύση. Ε, πρέπει οι κυβερνήσει μας επιπλέον να δράσουν και να πάψουν να μιλούν. Σκιώδης των Πρασίνων είναι παρόν, παρούσα. Μάλιστα. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο και ευχαριστώ πολύ για την συμβολή που υπήρξε γιατί από τη δική μας πλευρά θεωρούμε πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να, να, να καταπολεμηθεί η αδήλωτη εργασία και πιστεύω επίσης ότι ε, από, το τι, την πλευρά του τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια συντονισμένη προσέγγιση δεν θα ωφελήσει μόνο χώρες όπου το πρόβλημα είναι πραγματικά μεγάλο αλλά θα ωφελήσει και χώρες, όλες μάλλον τις χώρες της Ένωσης διότι η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας θα είναι όφελος για όλους. Θα πρέπει να ενισχυθεί ε, και μάλιστα θα ενισχυθεί, θα βελτιωθεί η κοινωνική και οικονομική κατάσταση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Υπάρχουν πολύ σημαντικέ παρατηρήσεις που ήδη έγιναν. Εγώ θέλω απλά να τονίσω κάτι ακόμα, ε, ότι πρέπει δηλαδή να προσέξουμε πάρα πολύ να μην χρησιμοποιήσουμε την αδήλωτη εργασία ώστε να υποστηρίξουμε την μείωση των ισχυωσών προδιαγραφών εργασίας ε, όπως συχνά γίνεται στις αγορές εργασίας γιατί πιστεύω πως στο παρελθόν έχουμε δει ιδιαίτερα σε χώρες όπου υπάρχουν αποτελεσματικά συστήματα πρόνοιας και υγειονομική ε, περιθάλψη ε, σταθερές οικονομίες το πρόβλημα είναι μικρότερο. Ε, δεν μπορεί δηλαδή ε, η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας να σημάνει ε, μείωση των προδιαγραφών απασχόλησης. Υπ' αυτή την προϋπόθεση έχω να κάνω και μια ερώτηση γιατί δηλώθηκε ήδη στις αρχές αλλά μόνο πολύ σύντομα ότι βέβαια η κρίση είχε ιδιαίτερη επιρροή στην κατάσταση της Αγοράσω ω προς την αδήλωτη εργασία. σω η κυρία Γκριν λοιπόν θα μπορούσε κάπω περισσότερο να το σχολιάσει. Ποιο είδο επιρροή υπήρξε από την κρίση, υπήρξε αύξηση τη αδήλωτη εργασία, τι μπορεί να γίνει για να καταπολεμηθεί αυτό το φαινόμενο και τέλο υπόθηκε ότι οι πιο ευάλωτε ομάδε είναι αυτέ που επηρεάζονται από την αδήλωτη εργασία. Μιλήσατε για πρόληψη πολύ. Τι μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένα για να προστατεύσουμε αυτές τις ομάδες. Μιλάω για τους άνεργους, για τους νέους και πώς αυτό μπορεί να ενσωματωθεί στην προσέγγιση πρόληψης που προσπαθούμε να θέσουμε σε εφαρμογή με αυτή την πλατφόρμα. Μάλιστα, υπάρχει κάποιο σκιώδης που δεν μπόρεσε να πάρει το λόγο. Τώρα πρέπει λοιπόν να σταματήσουμε γιατί μπορείτε τώρα να απαντήσετε για δυο 3 λεπτά για αυτά όλα τα ερωτήματα γιατί μετά ο χρόνος μας τελειώνει. Παρακαλώ, αν μπορείτε να μας κάνετε τουλάχιστον κάποια σχόλια για τα ερωτήματα που τέθηκαν. Μάλιστα, δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα, αλλά πολύ ευχαρίστως να διαβιβάσω πιο λεπτομερείς απαντήσεις γραπτός αργότερα. Όπως γνωρίζετε, η πρόταση της Κομισιόν είναι επιτάπητος, είναι υποσυζήτηση, αλλά το Συμβούλιο έχει προχωρήσει. Μια γενική προσέγγιση επετέφθη στη διάρκεια της Ιταλικής Προεδρίας πριν από κάποιες εβδομάδες και για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην πλατφόρμα τώρα Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τον εισηγητή και το Ευρωκοινοβούλιο για να μπορέσουν να ξεκινήσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα οι σχετικές δραστηριότητε μέσα στο 2015. Τώρα λοιπόν με το Συμβούλιο, με τη βοήθεια φυσικά της, Κομισιό... φυσικά της Κομισιόν που θα έρθει να συζητήσει τις διάφορες διατάξεις πιο συγκεκριμένα, πιο λεπτομερώς θα προχωρήσουμε. Για τον ορισμό, πιστεύω πως δεν πρέπει να κρύβουμε πως υπάρχει συζήτηση όντως και ότι ελπίζουμε πως η πλατφόρμα θα μπορέσει να βοηθήσει να προχωρήσουμε. Εμείς θέσαμε μια βάση αφετηρίας, όπως υπέδειξε και κάποιος ευρωβουλευτής, κυρίως βρίσκεται, υπάρχει για να εξασφαλίσει ότι δεν δουλεύουμε για παράνομη ε, δραστηριότητα όπως ε, ε, μπόριο ναρκωτικών ή ξέπλυμα χρήματο αν και σε ορισμένες περιπτώσεις, ορισμένες μορφές αδίλωτη εργασία μπορεί να συνδέονται και με μορφέ εγκληματικότητα. Όμω, πρέπει να εξακολουθήσουμε τη δουλειά με τα κράτη-μέλη λαμβάνοντας υπόψη, και αυτό το θέλω πολύ να το διευκρινίσω, ότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πως υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη, διαφορετικές εμπειρίες, διαφορετικά πλαίσια και ότι θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να συνεργαζόμαστε με τους εμπειρογνώμονες και τα κράτη-μέλη για να ορίσουμε καλύτερα τη μη δηλωμένη εργασία. Και αυτό προτείναμε ως δραστηριότητα της πλατφόρμας για να προχωρήσουμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο στη στρατηγική μας και στη δράση μας. Πιστεύουμε πως χρειάζεται συμμετοχή όλων των κρατών μελών, πράγμα το οποίο θα είναι η διαφορά σε σχέση με άλλες προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως τις διαφορές. Ωστόσο αυτό δεν εμποδίζει η ίδια η πλατφόρμα να μπορέσει να ορίσει τις προτεραιότητες αυτού του προγράμματος εργασίας και να υπάρξουν κάποιες δραστηριότητες που πάντως στην αρχή θα εφαρμοστούν με ομάδες των μελών, με κάποιους εμπειρογνώμονες πριν να διευρυνθούν σε όλα τα κράτη-μέλη. Για το θέμα των στόχων της πρωτοβουλίας αναφέρονται στην πρότασή μας. Πρόκειται για καλύτερη, την καλύτερη εφαρμογή του εθνικού δικαίου και του ευρωπαϊκού δικαίου για την ε, ε, ε, ύπαρξη θέσεων απασχόλησης ποιοτικές και δηλωμένες και βελτίωση της συνεργασίας ανάμεσα στις διάφορες αρχές των κρατών μελών, βελτίωση της τεχνικής δυνατότητας για κάλυψη των φαινομένων ε, διασυνοριακών μη δηλωμένων εργαζόμενων και βεβαίως ε, αύξηση ε, και πίεση για στα κρατημέλη ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε την αδήλωτη εργασία. Για τις λεπτομέρειες θα μπορούσα να επανέλθω με άλλη ευκαιρία, στα επόμενη ευκαιρία. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν νομίζω ότι έχουμε χρόνο γιατί δεν θα έχουμε και πολύ παραπάνω μαζί μας τους Ιερμηνείς. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στο πάνελ και για όλες τις ερωτήσεις που ακούσαμε. Για τα μέλη της Επιτροπής, ευχαριστώ. Παρά το γεγονός ότι δεν μπορέσαμε να ακούσουμε πάρα πολλές ερωτήσεις. Και θα θέλαμε να ξέρουμε λοιπόν ε, την άποψή σα για την αδελφή Όπω ξέρετε, θα συνεχιστούν οι εργασίε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να είναι τελικά καλή η έκθεση για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ λοιπόν ε, όλους του συμμετέχοντε, ευχαριστώ το πάνελ, ευχαριστώ και για όλε τι ερωτήσει που παρουσιάσατε εδώ πέρα στην Επιτροπή και πολύ λυπάμαι που δεν μπορέσατε όλοι σας να πάρετε το λόγο. Θα συνεχίσουμε το απόγευμα της συνεδρίασή μας με τις συζητήσεις με νέα πάνελ. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος.